Καλημέρα σας. Να καλωσορίσω το ακροτήριο τα μέλη της Επιτροπής ε, στη σημερινή συνεδρίαση. Όπως ξέρετε έχουμε μια ακρόαση ε, με τίτλο «Καταπολέμηση του ξεπλήματος παράνομων, ε, της νομιμοποίησης δηλαδή παράνομων προσόδων». στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Στο πρώτο πάνελ μας ε, θα μιλήσουμε για τους κινδύνους ε, για το ξέπλυμα ε, χρήματος μέσα στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό τομέα. Χρειαζόμαστε βοήθεια από επαγγελματίες φρουρούς Επίσης, ε, ε, σύμφωνα με τις τελευταίες, ε, τα τελευταία στοιχεία της Europol, μέχρι το 1,2 του ετησίου ευρωπαϊκού ΑΕΠ ε, εντοπίζεται ότι ε, συμμετέχει σε παράνομες ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Και αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά εκατομμύρια το χρόνο για τη συμμόρφωση προς το, το νόμο, καλύπτει μόνο το 1%. Μάλλον, συλλαμβάνει μόνο το 1% των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Το πρώτο τμήμα λοιπόν θα αφιερωθεί στην εξέταση των κινδύνων του χρήματος στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα μέσω επιλεγμένων παραδειγμάτων ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που πρόσφατα έχουν ε, δημιουργήσει ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος όπως η ABLB, η Τράπεζα της ε, Λετωνίας, η η Πιλάτος Μπάνκα στην Μάλτα και η ε, ε, Τράπεζα της Εστονίας. Ε, ορισμένοι λένε ότι στοχεύονται οι μικρότερες χώρες που μπορεί να ξεπεραστούν από το έργο ε, της παρακολούθησης των, ε, του τραπεζικού του τομέα αυτό θα δούμε αν δικαιολογείται. Για να μην σας δώσω όμως ε, μόνο αρνητικά νέα, θα σας θυμίσω την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο, δηλαδή άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες των τραπεζικών λογαριασμών προς τις αρχές επιβολής του νόμου θα είναι ένα ακόμα βήμα στην καταπολέμηση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Για αυτό το πρώτο πάνελ έχουμε καλέσει εκπροσώπους από τα διάφορα εποπτικά ε, ε, όργανα που θα μας δώσουν πληροφορίες από πρώτο χέρι για αυτές τις περιπτώσεις, για αυτές τις υποθέσεις μάλλον. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την παρουσία του σήμερα εδώ. Θα ήταν καλό να είχαμε και εκπροσώπους των ιδίων των τραπεζών που αναμεγνύονται σε αυτά τα περιστατικά, αλλά δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό. Είτε λόγω ε, ηλυμένων υποχρεώσεων των εκπροσώπων τους, είτε επειδή δεν ήταν πλήρης η συμβολή τους ή μπορεί να ήταν πρώιμη, πρώιμο στάδιο, γιατί υπάρχουν, είναι ακόμα στα δικαστήρια οι συντονιστέ τη επιτροπή μετά από αυτή την ακρόαση μπορεί να αποφασίσουν να κάνουν μια μεταγενέστερη ακρόαση με τι τράπεζε που έχουν δημιουργήσει ανησυχίε ω προ το ξέβλημα χρήματο. Επίση, ο κ. Ζαμάλα Ελχίντη, που είναι ε, ε, αναπληρωτής διευθυντής ε, του δικτύου οικονομικών εγκλημάτων του, ΙΠΑ, του ΦΙΝΣΕΝ, ε, δεν μπόρεσε να δεχτεί την πρόσκλησή μας. Ε, έχει όμως στείλει μία συγκεκριμένη πρόταση για νομοθεσία ε, για την τράπεζα EBLV. Εξάλλου θα έχουμε επαφές μαζί του τον Ιούλιο που θα πάμε στη Ουάσιγκτον. Το δεύτερο πάνελ θα αφιερωθεί ε, στην αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι σε, ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι για ξέπλυμα χρήματος. Όλα τα μέλη έχουν λάβει ε, τις γραπτές απαντήσεις ε, των εισηγητών στα ερωτήματα που τους στείλαμε πριν από την ακρόαση αυτή και απαντήσεις αυτές υπάρχουν και στο δίκτυο. Ε, στο website της Επιτροπής μας. Η μέθοδος εργασίας για τα δύο πάνελ θα είναι η εξής. Κάθε ομιλητή θα έχει μάξιμο με 7 λεπτά για εισαγωγικέ παρατηρήσει. Μετά από την παρουσίαση των ομιλητών, την εισήγηση μάλλον του κάθε ομιλητή, θα υπάρξει μια συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Οι ερωτήσεις θα τεθούν σε χρονοθυρίδες πεντάλεπτες ένα λεπτό η ερώτηση και ο υπόλοιπο χρόνο αφιερωμένο στην απάντηση. Αν ο χρόνο το επιτρέπει, ο βουλευτή θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει υπερώτηση χωρί να ξεπεράσει το πεντάλεπτό του. Θα σας παρουσιάσω τώρα τους ομιλητές του πρώτου πάνελ που είναι ο κύριος Πέτερ Πουτνίν πρόεδρος ε, της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής και Κεφαλαιακής Αγοράς ε, της ε, Λετωνίας που θα μας μιλήσει για την υπόθεση ABLV. Έπειτα έχουμε την κυρία Μαριάννη Σικλούνα, Γενική Διευθύντρια της Μαλτέζικης Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, τον κύριο Κένεθ Φαρούτζα, που είναι Διευθυντής της Μαλτέζικης Υπηρεσίας ε, Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών θα μας δώσει πληροφορίες για την ε, Τράπεζα Πιλάτους και έχουμε και τον κύριο Αντρέ Μόμ που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ε, Αρχής Δημοσιονομικής Εποπτείας και Εξυγίανσης και που θα μας διαφωτίσει για τις υποθέσεις της Danske Bank και της Verso Bank. Ο κύριος Πούτνινς πρώτα λοιπόν θα κάνει την εισήγηση του excuse Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να σας μιλήσω εδώ για θέματα καταπολέμησης της νομοποίησης παράνομων εσόδων ε, στην Λετωνία και ιδιαίτερα για την τράπεζα APLV. Θα δείτε μια σύντομη παρουσίαση στις οθόνες σας και θα προσπαθήσω στα πέντε λεπτά που μου δίνετε να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία. Καταρχάς το γενικό πλαίσιο. Ο συνολικός αριθμός εμπορικών τραπεζών ε, στην ε, Λετωνία είναι 16. Αν αφαιρέσουμε την ABLV ε, είναι 15. Τρεις από αυτές είναι τράπεζες λιανικής για τους εγχώριους πελάτες, ενώ 12 είναι τράπεζες για αλλοδαπούς όπως τις λέμε, που εξυπηρετούν κυρίως αλλοδαπούς ε, πελάτες. Η παρουσία μεγάλου αριθμού αλλοδαπών πελατών, ιδιαίτερα από την Ανατολική Ευρώπη, πάντα ήταν ε, σημαντική πρόκληση και παράγοντας κινδύνου για την εποπτεία των τραπεζών στη Λετωνία ήδη από τη δεκαετία του 1990 και γι' αυτό το FCMC έχει ζητήσει από τις ε, τράπεζες να, αυξήσουν, ε, τις, να ε, εφαρμόζουν αυξημένες απαιτήσει, όπως για παράδειγμα ο, ο, λόγος κεφαλαίου υποχρεώσεων, η, ο δείκτης ρευστότητας κλπ. Τώρα πρέπει να κάνουν σημαντική αναθεώρηση η Λετωνία και να επεξετάσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα που έχουν αποδειχθεί μη βιώσιμα. Όσον αφορά την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων, το επίπεδο καταθέσεων της αλλοδαπής ε, έφτασε ε, στο υψηλότερο σημείο το 2015, σχεδόν το 55% των συνολικών καταθέσεων στη Λετωνία. Μετά από την ε, σύσφυξη των ε, διεθνών προτύπων και την προσχώρηση της Λετωνίας ε, στον ΩΣΑ το 2016 έχει αλλάξει η εποπτική προσέγγιση και τώρα η FCMC ζητάει από τις τράπεζες να επανεξετάσουν τους πελάτες τους και να αποφύγουν χρήματα αμφίβολης προέλευσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείωση των ε, ανωδοπών καταθέσεων, έχουμε φτάσει στο 31% τώρα πια ήδη και εξαιρώντας την τράπεζα ABLV ε, πλησιάζουμε το κατόφλι του 20% που πιστεύουμε ότι θα το φτάσουμε σε 3-4 μήνες. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο καταθέσεων της αλλοδαπής σε τα τελευταία 20 χρόνια και οι προσπάθειες ε, θα συνεχιστούν. Διότι ε, αυτό είναι κάτι που επιβαρύνει την φήμη των τραπεζών μας ε, στο εξωτερικό. Επιπλέον έχει αλλάξει η πολιτική κατάσταση στον κόσμο σήμερα. Ε, και η Λετωνία και άλλα κράτη της ε, Βαλτικής ε, βλέπουν ότι έχει αλλάξει η κατάσταση και η θέση της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να μειώσουμε όσο γίνεται το ποσοστό ξένων καταθέσεων και να φτάσει στο 5% των συνολικών καταθέσεων. Λίγα λόγια για τις κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει η FCMC. Ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι τράπεζες θα πρέπει να συνάδει με το σύστημα ελέγχου τους ε, καθώς και με τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Εάν υπάρχουν σημαντικές τροποποίησεις ε, στους εθνικούς στις εθνικές ε, ρυθμίσεις, στους εθνικούς κανόνες, θα πρέπει να φροντίζει ο νομοθέτης ε, για την ε, εφαρμογή τους και οι τράπεζες θα πρέπει να περνούν σε πελάτες χαμηλού κινδύνου. Η Λετωνία στηρίζει αυτή την προσέγγιση και η FCMC έχει εποπτεύσει ιδιαίτερα αυστηρά την τράπεζα ABLV. Συνεχίζει η Λετωνία να ε, αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την ε, νομοποίηση παράνομων ε, εσόδων, αλλά έχουν ενταθεί προσπάθειες της FCMC τα τελευταία δύο χρόνια. Όλοι ξέρουμε ότι το 2016 επιβλήθηκε πρόστιμο στην ABLV, το υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ σε τράπεζα της Λετωνίας. Επίσης ε, εξετάστηκε η τράπεζα όσον αφορά ε, θέματα της Βόρειας Κορέας πέρσι και ε, λάβαμε διορθωτικά μέτρα για να μειώσουμε την έκθεση της τράπεζας αυτής και περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ στήχησε η προσπάθεια αυτή. Όλα αυτά είναι άνευ προηγουμένου στην Λετωνία και θα πρέπει να πω ότι οι περισσότερες κατηγορίες που ε, δημοσιεύτηκαν σε σχέση με την ABLV ε, δεν ε, απευθύνονταν στην FCMC. Μάλιστα τα περισσότερα από τα θέματα που αναφέρθηκαν σε αυτό το δημοσίευμα ήταν πράγματα που εξετάζαμε ούτως ή άλλως και εγώ θεωρώ ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν, ότι το παρελθόν ε, είχε παίξει τόσο αρνητικό ρόλο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα κλείσω εδώ και ευχαρίστω θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Βλέπω ότι ήδη έλειξε ο χρόνος μου. Σας ευχαριστώ. Uh, Well, now Σας ευχαριστώ πολύ και από το βορρά πάμε στο νότο. Πράγμα που σημαίνει ίσως ότι τα θέματα που συζητάμε σίγουρα δεν έχουν να κάνουν με περιφέρειες. Δεν είναι τοπικά. Γι' αυτό θα ε, δώσω λοιπόν το λόγο στην ε, κυρία Μαρία Σικρούνα που είναι Γενική Διευθύντρια της ε, Υπηρεσίας Χρηματοπιστωτικού ε, της ε, αρχής μάλλον ε, χρηματοπιστωτικού ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα να πάρω το λόγο. Ε, τώρα, ε, ε χρόνο, θα, σας, θα αναφέρω κάποια από τα κομμάτια της γραπτής εισήγησης που σας έχω στείλει. Η γραπτή εισήγηση σας έχει σταλεί και μπορείτε να την ε, μελετήσετε. Έχουμε διάφορες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε σε, στην περιπόθεση της Τράπεζας Πιλάτους. Εμείς συγχαίρουμε την πρωτοβουλία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, το, κανόνες που θα επιβάλλουν στις ε, τοπικές ρυθμίσεις να ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όπως και ε, σε άλλες περιπτώσεις ακολουθήσαμε αυτήν την πορεία και για την υπόθεση του πιλότου Έχουμε ε, βάλει διάφορα θέματα, διάφορες πληροφορίες. Ε, στείλαμε τις ε, πληροφορίες που ζητήθηκαν και επίσης αναθέσαμε ε, σε τρίτο ανεξάρτητο μέρος την διενέργεια αυτής της έρευνας. Και μετά από πάνω από 12 μήνες επιτρέψαμε στην τράπεζα και εδώ ήθελα να τονίσω ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία και οι προθεσμίες αδειοθότησης. Έκτοτε η Τράπεζα Πιλάτους ε, έχει υποστεί ψηλό βαθμό εποπτείας. Έχουμε την ε, ε, επιβολή FIU, την εποπτεία τη δέουσα επιμέλεια και διαρκώς μας έδινε τις απαραίτητες δηλώσεις. Η εποπτική έκθεση για διάφορες πτυχές ε, εντατικοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια όταν διέρευσαν οι διάφορες καταγγελίες και στα ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης εναντίον αυτής της τράπεζας. Και ε, με την FCA ακολουθήσαμε όλη την προβλεπόμενη διαδικασία. Με βάση τις πληροφορίες που είχαμε συγκεντρώσει παλαιότερα αλλά και στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου ξεκινήσαμε μια συνολική και εις βάθος ε, εξέταση της ε, τράπεζας μαζί με την AIU. Εξετάσαμε όλους τους λογαριασμούς, τις συναλλαγές, τη διακυβέρνηση, για να έχουμε μια γενική εικόνα και να έχουμε και μια στεναρή αξιολόγηση για το κατά πόσο η τράπεζα αυτή είχε αναμειχθεί σε ξέπλυμα χρήματος. Αυτή η εξέταση εξακολουθεί. Και σε αυτή την περίπτωση οι ε, βασικές πληροφορίες που είχαμε είναι οι, προληπτικοί δείκτες που, δίνονται στους ρυθμιστές με συγκεκριμένους δείκτες, αλλά βέβαια ε, είναι σχετικά περιορισμένη. Επιπλέον, η δέουσα επιμέλεια, όσο και αν προσπαθούμε να είναι συνολική και καθολική, από μόνη της περιορίζεται γιατί οι ρυθμιστές δεν έχουν απαραίτητο στην πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές ε, επιβολής του νόμου. Όταν όμως ε, ε, μάθαμε την απόφαση των αρχών των ΙΠΑ να ε, διώξουν δικαστικά τους εκπροσώπους της τράπεζας αμέσως προβήκαμε στα απαραίτητα βήματα, αντικαταστάθηκε ο διοικητής και ε, ε, υποτέθηκαν υπό έλεγχο οι συναλλαγές της τράπεζας αυτής. Παρακολουθούμε λοιπόν την κατάσταση και αναλύουμε τα αποτελέσματα των εκθέσεων που έχουμε συγκεντρώσει για να αποφασίσουμε τι, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Ο ρόλος της UNFSA και μάλλον την MFSA είναι να ρυθμίσει την, και να ελέγξει τη συμπεριφορά των τραπεζών. Επιπλέον υπάρχει και η Μαλτέζικη Μονάδα Ανάλυσης ε, ε, Οικονομικών Συναλλαγών που συμπληρώνει την MFSA. Ε, Αυτά τα θέματα έχουν άμεσες επιπτώσεις στην προληπτική εποπτεία, όπως έχουμε δει ξεκάθαρα από τις υποθέσεις που έχουν ε, έρθει στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, ε, όπως και στην υπόθεση Πιλάτος. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ενισχύσει σημαντικά και δώσει νέα ε, έμφαση στα θέματα της καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος και στην ενίσχυση της εποπτείας το 2016. Η MFSA ε, σταθεροποίησε την μονάδα που προβαίνει στον ε, χρηματοπιστωτικό έλεγχο. Η, η ιδέα ήταν να έχουμε μια πιο κεντρική ομάδα εμπειρογνωμοσύνης. Μαζί με την FIU έχουμε εισάγει μια νέα μεθοδολογία με βάση τον κίνδυνο και συνεχίζουμε να ερευνούμε και να επεκτείνουμε και να βαθύνουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας ιδιαίτερα κεντρικό θέμα είναι η συνεργασία μεταξύ της εποπτείας και της προληπτικής εποπτείας, prudential έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ε, ε, ολοκληρωμένη εικόνα για τις υποθέσεις αυτές. Εξακολουθούμε να ωφελούμεθα από επιπλέον πόρους και επιπλέον κατάρτιση. Έχουμε μεταβεί στη ΣΥΠΑ για το λόγο αυτό και επίσης έχει υπάρξει και καλύτερο συντονισμός με τις αντίστοιχες ε, Αμερικανικές αρχές. Γι' αυτό και καλωσορίζουμε την ε, νέα στρατηγική ε, ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος που ξεκίνησε στην, ανακοινώθηκε στη Μάλτα πριν από λίγες εβδομάδες και στόχο έχει να, ενισχυθεί η συνεργασία των διαφόρων οργανισμών ιδιαίτερα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Θα χρειαστεί ε, ε, μάλλον πιστεύουμε πως θα ωφεληθούμε από τις νέες κατευθυντήριες γραμμές και τα πλαίσια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν τρεις κεντρικοί τομείς ε, όπου θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε. Η εξολόγηση των επιχειρηματικών μοντέλων προτύπων των τραπεζών, όπου δεν έχουμε από την ΕΟΦΗΝ συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό θα μπορούσε να είναι κίνδυνος από την πλευρά της, ε, την οπτική MML, MFD, θα έπρεπε να υπάρχουν πιο συγκεκριμένες ε, ε, κατευθύνσεις να δούμε ποια είναι ακριβώς η δομή, ποια είναι, ποιοι είναι οι μέτοχοι, γιατί κάτι τέτοιο θα, είναι, θα ήταν πολύτιμο ως πληροφορία. Επίσης, η δέουσα επιμέλεια και η παρακολούθηση δεν αναφέρονται στο σημερινό πλαίσιο. Νομίζω πως αν είχαμε κάποιες επιπλέον οδηγίες θα ήμασταν πιο σε καλύτερη θέση ε, ε, ε, εγώ ολοκληρώνω λέγοντας πως το ξέβλημα χρήματος είναι πολύ σημαντικό θέμα, είναι μια μεγάλη πρόκληση για ολόκληρη την Ευρώπη και επαναλαμβάνουμε την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε το ξέβλημα χρήματος για να προστατέψουμε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Όργανο ώστε το σύστημα να ενισχυθεί. Ευχαριστώ τον κυρία Σικλούνα. τώρα ο Διευθυντής ε, του ε, FIU της Εποπτικής Αρχής της Μάλτα. Ο κύριος Φαρούτζα. Θα είμαι συνοπτικός. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μας προσκαλέσατε σήμερα. έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα συστήματα μας, συστήματα καταπολέμησης, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Έχουμε δύο ε, βασικές λειτουργίες, είναι αναλυτικού τύπου εποπτικές λειτουργίες, αναλύουμε τον πιστοτικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τις υπόλοιπες ε, εποπτικές αρχές, συνεργαζόμαστε με τις ε, διοκτικές αρχές, είμαστε επίσης υπεύθυνοι για την εποπτεία ε, επιχειρήσεων όπως πιστοτικά ιδρύματα κτλ. Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους ε, έχουμε αρμοδιότητες, η προσπάθειά μας είναι δύσκολη σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει συνεχώς, ιδιαίτερα στον, στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το προσωπικό μας και αυτό αντικατοπτρίζει την αύξηση των δραστηριοτήτων μας. Η καταπολέμηση πάντως της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων ε, συνεχίζεται και μπορούμε να λειτουργήσουμε αναλυτικά εφόσον έχουμε στη διάθεσή μας ε, τις κατάλληλες ε, αρμοδιότητες και τους κατάλληλους μηχανισμούς. Τα φαινόμενα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι αυστηρά εθνικά, είναι διασύνοριακά όλες οι χώρες προσπαθούν να συνεργαστούν στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος σε διεθνές επίπεδο και εκεί ο ρόλος μας είναι σημαντικός. Κάνουμε τακτικές αξιολογήσεις οι οποίες θεωρούνται χρήσιμες αλλά δεν αρκούν φυσικά. Πιστεύουμε ότι οι αξιολογήσεις και η μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιούμε θα μας βοηθήσουν να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Εν τω μεταξύ οι αξιολογήσεις οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί στα πλαίσια της αναθεωρημένης μεθοδολογίας δείχνουν ότι πάνω από τις μισές χώρες μέλη που αξιολογήθηκαν έχουν πετύχει αποτελέσματα μεσαίου ή ελαφρά ανώτερα από μεσαίο επίπεδο. πάντως τώρα πλέον ε, διώκονται και πολλές φορές καταλήγουν στην καταδίκη αυτών που συμμετέχουν στα δίκτυα νομιμοποίησης. Έχουμε και εμείς εθνικές μεμονωμένες εμπειρίες και πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει ε, να συνεχιστεί, την οποία έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα σε σχέση με την ε, δραστηριότητα την εποπτική. Έχει ξεκινήσει επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλαπλές νομοθετικές ρυθμίσεις για, την βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Ιδιαίτερα σε τομείς τους οποίους η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι περιορισμένη. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να ξεπεράσουν την πρακτική ε, δραστηριοποίησή τους στον τομέα αυτό ε, απομονωμένοι από τις υπόλοιπες χώρες γιατί σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα των προσπάθειών τους δεν διαδίδονται όπως θα έπρεπε. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσει προληπτικά και να παρέχει την τεχνική συνδρομή και την καθοδήγηση για την εφαρμογή των νέων κανόνων. Οι ευρωπαϊκές αρχές φυσικά είναι δραστήριες στον τομέα αυτό, αλλά καλύπτουν μόνο τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ε, δεν καλύπτονται οι μη χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και τα μη χρηματοπιστωτικά επαγγέλματα. Σχετικά τώρα με την νομοθεσία, πιστεύουμε ότι επειδή οι εξελίξεις είναι ταχύτατες θα πρέπει και οι νομοθετικές ρυθμίσεις να ακολουθούν τις εξελίξεις και να τις προλαμβάνουν. Θα πρέπει να προβλέπουμε σωστό χρονισμό για την υιοθέτηση των μέτρων τα οποία λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, αυτό το οποίο εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό είναι η συλλογή πληροφοριών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών. Εδώ έχει μεγάλη σημασία για μια ακόμη φορά η συνεργασία ανάμεσα στις εποπτικές αρχές. Σε επίπεδο διερεύνησης ανακρίσεων ε, δικαστικών διαδικασιών, ε, η συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Πολλές φορές ε, οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται σε μία, από μία εποπτική αρχή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δίωξη και τελικά τον βασικό στόχο που είναι η κατάσχεση των παρανόμων αυτών αποκτηθέντων εσόδων. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Αντρέ Νόμ, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ε, Αρχής της Εστονίας ε, για την χρηματοοικονομική εποπτεία. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που μας δίνατε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τα τελευταία αποτελέσματα της αρχής μας ε, και ε, τις προοπτικές όσον αφορά τον κίνδυνο. Έχουμε κάποιους κανόνες περί εμπιστευτικότητας. Νομίζω όμως παρόλα αυτά ότι μπορώ να σας δώσω αρκετά αναλυτικά στοιχεία. Η Finance Inspection είναι η αρχή χρηματοοικονομικής εποπτείας της Εστονίας. Εποπτεύουμε τα πιστοτικά ιδρύματα, τα, τις διαδικασίες τους, ε, έχουμε ελέγχους και συστήματα για να ε, προλάβουμε την ε, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την νομοποίηση παράνομων εσόδων. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ξεκίνησε τις εργασίες του το 2014. Ε, ήδη από την αρχή θεωρήσαμε ότι η καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων ε, και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελούσαν ε, σημαντική προτεραιότητα. Εισάγαμε νέα μοντέλα παρακολούθησης που βασίζονται στον κίνδυνο. Καταλαβαίνουμε τους ε, κινδύνους ε, και γι' αυτό ε, έχουμε αυξημένες εποπτικές δράσεις. Και ήδη το 2014 διαπιστώσαμε ότι δύο τράπεζες ήταν τράπεζες υψηλού κινδύνου. Η Δανέζικη τράπεζα Danske Bank που δραστηριοποιούταν και συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην Εστονία με βάση την ελευθερία της εγκατάστασης και ε, μια κάπως μικρότερη τράπεζα ε, με σε τους πολίτες της Ουκρανίας. Θέλαμε λοιπόν ε, να στείλουμε σαφές μήνυμα ότι η ιστορία δεν είναι ο κατάλληλος τόπος για μη διαφανείς ενέργειες και αυτό αφαιρέσαμε την άδεια των τραπεζών αυτών. Εδώ βλέπετε κάποια αριθμητικά στοιχεία ε, σχετικά με τις αυξημένες εποπτικές μας δράσεις ε, και εδώ έχουμε τα στοιχεία ε, από το 2014. Φαίνεται εδώ η εξέλιξη όσον αφορά τα, τις καταθέσεις αλλοδαπών. ξεκινήσαμε από σχεδόν 20% ενώ τώρα έχουμε φτάσει σχεδόν στο 11%. Ε, και αν συμπεριλάβουμε και τις offshore, ε, ξεκίνησαμε από 8,5% και έχουμε φτάσει σχεδόν, ε, και έχουμε φτάσει λιγότερο από 1,5%. Η κίνδυνη, λοιπόν στην Εστονία είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι ήταν το 2014 που ξεκινήσαμε αυτήν την πιο επιθετική εποπτεία. Εδώ βλέπετε στατιστικές εξωτερικών πληρωμών στην Εστονία και αυτά, τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τον κίνδυνο για νομοποίηση παράνομων εσόδων. Βλέπετε ότι οι πληρωμές από την Εστονία έχουν μειωθεί πολύ. Από 31 δισεκατομμύρια ευρώ σε 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να είμαστε σαφείς λοιπόν, η εποπτεία για την αποφυγή της νομοποίησης παράνομων εσόδων ε, συνεχίζεται. Έχουμε δεσμευτεί να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και νομίζω ότι στέλνουμε πια το μήνυμα ότι η Εστονία δεν είναι το κατάλληλο μέρος ε, για ε, νομοποίηση παράνομων εσόδων ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νόμε, ευχαριστώ ε, η χρηματοδοτηση Νήμε, ευχαριστώ και σας ευχαριστω ευχαριστω πολυ κυριε νομε ευχαριστω και ολους τους ομιλητες θα ξεκινησει τωρα η συζητηση με τους ευρωβουλευτές. Ένα λεπτό η καθερώτηση, τέσσερα λεπτά για την απάντηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις που ακούσαμε και καθότι ασχολούμαστε με συγκεκριμένες ε, υποθέσεις, ε, θα ήθελα να επικεντρωθώ ε, στην Danske Bank και τη Bank. Κύριε Αντρενόμ, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις, λοιπόν, προς εσάς. Οι δανέζικες αρχές πότε ενημερώθηκαν ε, πρώτη φορά ότι μια μεγάλη τράπεζα εντός του εδάφους τους ε, ήταν ε, ύποπτη για καταπολέμηση παράνομων εσόδων στην Εστονία. Πότε και πώς ενημερώθηκαν και τι απάντηση λάβατε και τι δράσεις αναλάβατε μετά. Σε άρθρο δανέζικης εφημερίδας ε, λέει ότι οι εστονικές ε, ότι οι ε, αρχές φοβήθηκαν ότι λαμβάνουν παραπλανητικές πληροφορίες από τις δανέζικες αρχές. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι παραπλανητικές πληροφορίες. Θα επανέλθουμε μετά στις ε, απαντήσεις. Θα κλείσω εδώ την πρώτη μου ερώτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόμ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, όπως σας είπα, ήδη το 2014 πήγαμε στην Τάνσκε και είχαμε επιτέλους ε, επιθεώρηση ενημερώσαμε την ε, Δανέζικη Εποπτική Αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα. Καλύψαμε ε, επίσης την Danske Bank ε, στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας με μια ανάλυση τύπου ΣΡΕΠ διότι θεωρήσαμε ότι είναι υπερβολικά υψηλός ο κίνδυνος. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τις δανέζικες αρχές. Διεξάγαμε την εποπτική μας ανάλυση στην Εστονία και ήταν πολύ σαφής ο στόχος μας. Ε, άλλωστε έχει σταματήσει τις ε, δραστηριότητε αυτές η τράπεζα στην Εστονία. Για μας ως εποπτική αρχή είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Για την Εστονία τα πράγματα είναι απλά. Εάν Ο βασικός μας στόχος είναι να σταματήσουν αυτές οι δραστηριότητε στην Εστονία. Να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας ευθέω. Ναι, φυσικά ε, όλο αυτό το διάστημα Καθ' όλη τη διάρκεια της περίπτωση αυτής, της υπόθεσης αυτής, είχαμε επαφές με τις δανέζικες αρχές. Και είχατε μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τις παραπλανητικές πληροφορίες. Νομίζω ότι αναφέρεσα στο γεγονός ότι το άρθρο στην εφημερίδα και ανέφερε ότι εντός της Danske Bank ήταν κάτι γνωστό, ότι υπάρχει δηλαδή μεγάλος κίνδυνος νομοποίησης παράνομων εσόδων στην Εστονία και ότι υπήρχε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος από την Ρωσία. Εμείς ήδη το 2014 κάναμε επιτόπου επιθεώρηση και η Danske Bank δεν μας είχε ενημερώσει για τις υποψίες που είχαν για κάποιους πελάτες. Τώρα όμως ε, έχουμε, είμαστε σε επαφή με τις ε, δανέζικες ε, αρχές και είχαμε ε, στείλει όλε τι πληροφορίε που είχαμε λάβει. Δεν μπορώ να σα πω περισσότερο γιατί είναι ακόμα μια ανοιχτή υπόθεση αυτή. Σα ευχαριστώ για την ε, απάντηση αυτή, αλλά μου φαίνεται ότι η συνεργασία ανάμεσα στι Δανέζικε και τι Εστονικέ Αρχέ δεν είναι σαφές για μένα αν είναι αποτελεσματική και τι ε, δράσεις έχουν αναλυφθεί. Ξέρω ότι είναι ακόμα μια ανοιχτή υπόθεση, αλλά νομίζω ότι μας δείχνει μια από τις αδυναμίες που έχουμε στη συνεργασία μεταξύ αρμοδίων αρχών. Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας. Οι εστονικές αρχές έκαναν κάτι από μόνες τους ή απλά ενημέρωσαν τις δανέζικες αρχές και πώς ήταν η συνεργασία μεταξύ των αρχών. Ναι, φυσικά τα πάντα κάναμε. Ήδη το 2014, όπως σας είπα, ε, είχαμε, διενεργήσαμε επιτόπου επιθεώρηση, ήμασταν ε, ικανοποιημένοι. Ε, ζητήσαμε από την Danske Bank να αλλάξει η επιχειρηματική στρατηγική και να σταματήσει τις, ε, τις δουλειές της με αλλοδαπούς. Η Danske Bank ε, αντέδρασε και σταμάτησε τις δραστηριότητες αυτές στην Εστονία. Να σας εξηγήσω όμως πώς έχει το θέμα των ευθυνών μεταξύ των εποπτικών αρχών. Η Danske Bank υποφελήθηκε ε, του δικαιώματος ε, της ελεύθερης εγκατάστασης στην Εστονία. Εμείς ε, ως αρχή εποπτεύουμε θέματα νομοποίησης παράνομων εσόδων. Κάποια θέματα διακυβέρνησης όμως είναι ακόμα στα χέρια της αρχή της ε, έδρα ε, της τράπεζας. Νομίζω ότι είχαμε καλή συνεργασία με τις δανέζικες αρχές. Επικεντρωθήκαμε στα θέματα νομοποίησης παράνομων εσόδων. Λύσαμε το θέμα όσον αφορά την Εστονία. Και τώρα πια οι δανέζικες αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να κάνουν κάτι σε επίπεδο διακυβέρνησης. Νομίζω όμως ότι ήταν εξαιρετική η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρχές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τη θέλει διευκρίνηση. Παρακαλώ όμως να προσπαθήσουμε να περιοριστούμε στα πέντε λεπτά συνολικά ανά ομιλητή. Ο κύριος Κάρινς από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θέλω να ευχαριστήσω τους, δύο, τους τρεις ομιλητές θέλω να στρέψω την προσοχή μου στην περίπτωση της ABLV στη Λετωνία, στη δική μου χώρα. Η ερώτησή μου αφορά δηλαδή τον κύριο Πούτνιτς και θα ομιλήσω τη Λετωνική γιατί είναι περίεργο δύο Λετωνοί να ομιλούν μεταξύ τους ξένη γλώσσα. Αν ε, ενθυμίστε, εμείς εδώ ο ρόλος μας είναι νομοθετικός, είμαστε συνομοθέτες. Ο έλεγχος των πιστοτικών ιδρυμάτων ε, βρίσκεται στις εποπτικές αρχές της κάθε χώρας και στην Λετωνία στη δική σας οργάνωση, στο δικό σας οργανισμό. Εγώ άκουσα την παρουσίασή σας σήμερα, το... έχω σημειώσει και τις απαντήσεις γενικά που έχετε δώσει μέχρι τώρα και η αίσθησή μου είναι ότι όλα πάνε καλά, ε, όλα είναι εντάξει, όλα λειτουργούν με το σωστό τρόπο. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξής. Αν όλα πράγματι πάνε καλά, πώς είναι δυνατόν μια τέτοια περίπτωση της ABVLB ε, να συμβεί. Μιλάμε για ένα οικονομικό έγκλημα. Είναι κάτι το οποίο θέτει σε αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων σας, των εργασιών σας. Αν πράγματι ασκείτε μια σωστή εποπτεία, γιατί συνέβη αυτό το οποίο συνέβη και γιατί η πληροφόρηση δεν έγινε από την υπηρεσία σας ή από άλλες εποπτικές αρχές, αλλά ήρθε από το Φίνσεν των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν έχουμε να κάνουμε σαφώς με αρκετές ελλείψεις σε επίπεδο ε, συνεργασίας. εφόσον ελέγχετε ε, τις μεγάλες τράπεζες να μην σας διαφεύγουν κάποιες άλλες. Λοιπόν, μπορείτε να δώσετε κύριε Πούτνιτ την απάντησή σας. Όπως είπα προηγουμένως, τα στοιχεία τα οποία έδωσε το Φίνσεν ήσαν γνωστά στην εποπτική αρχή και τα στοιχεία που έστειλε το Φίνσεν εμείς του τα δώσαμε. Τώρα γιατί συνέβη αυτό. Δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπος του Φίνσεν ήταν παρόν θα μπορούσε να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως είμαι πεπισμένος ότι τα στοιχεία αυτά τα οποία κυκλοφόρησαν αναφέρονται σε ε, παλαιότερους χρόνους. Είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αναφέρονται στη σχέση της συγκεκριμένης τράπεζας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικανικής κυβέρνησης τα οποία ακόμα είναι σε εκκρεμότητα. Πάντως εμείς όπως είπα και στην ομιλία μου βγάλαμε τα κατάλληλα συμπεράσματα δεν υπήρξαν ιδιαίτερες εκπλήξεις, συγγνώμη. Διακόπτει ο κύριος Κάρινς. Στα αγγλικά. Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι δεν μας έδωσε κάτι το καινούριο το Φίνσεν, κάτι που δεν το ξέραμε. Αλλά χάρη στην έκθεση Φίνσεντ η τράπεζα αυτή κλείνει τώρα. Γιατί δεν την είχατε κλείσει την τράπεζα εσείς νωρίτερα αν είχατε τις ίδιες πληροφορίες. Δεν έχει νόημα η στάση σας. Ή το ξέρατε και έπρεπε να την κλείσετε ή δεν το ξέρατε και τώρα που το μάθατε την κλείνετε. Σωστή η ερώτησή σας και νομίζω ότι θα σας δώσω την κατάλληλη απάντηση δεν έκλεισε την τράπεζα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ένα σχέδιο ε, εγγράφου Η τράπεζα αυτή τη στιγμή δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία αυτά ουσιαστικά ε, πτώχευσε μέσα σε τρεις-τέσσερις μέρες. αμφισβήτησαν οι Αμερικανικές υπηρεσίες ε, την ε, ικανότητα της τράπεζας να επιβιώσει μετά από τη δημοσίευση των στοιχείων αυτών. Όταν έρχονται από πλευράς του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών τέτοιου είδους στοιχεία και πληροφορίες ε, δεν μπορεί να επιβιώσει ένα πιστοτικό ίδρυμα. Ίσως πριν 10 χρόνια αυτό να ήταν εφικτό, αλλά τώρα πλέον δεν είναι εφικτό. Οι αγορές απομονώνουν την τράπεζα αυτή. και δεν έχει κανένα λόγο να προσφύγει σε διαδικασία πρόσβασης η συγκεκριμένη τράπεζα διότι έχει πλέον απομονωθεί πλήρως από τις αγορές. Είναι λοιπόν σε εκκρεμότητα οι δραστηριότητες οι τραπεζικές του συγκεκριμένου ιδρύματος και αν κάποια τράπεζα στην Ευρώπη επηρεαστεί από τέτοιου είδους έγγραφα, ταμιακά θα φύγει και δεν έχει καμία δυνατότητα επιβίωσης. Και αυτό που είπατε κλείσιμο της τράπεζας, το shutdown, στην ουσία αντικατοπτρίζει την αντίδραση των αγορών. Όχι ότι η Αμερικανική κυβέρνηση απέσυρε την άδεια λειτουργίας, αυτό είναι αρμοδιότητα αποκλειστική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Κάριν θα ήθελε ξανά το λόγο, αλλά δεν έχουμε πλέον χρόνο. Ε, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θα πάρουν το λόγο, η κυρία Γκόμες. προς τους εκπροσώπους των οργάνων της Μάλτα μετά τη δολοφονία ε, της δημοσιογράφου ε, σας κάναμε πάρα πολλές ερωτήσεις σε σχέση με τον ιδιοκτήτη της mm. τράπεζας Πιλάτους. Δεν είμαστε εμπειρογνώμονες, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά. Είπατε ότι πράγματι η τράπεζα αυτή είχε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Ε, γιατί δεν είχατε κλείσει την τράπεζα ή μάλλον γιατί δεν την έχετε κλείσει ακόμα. Τώρα για την εποπτική αρχή είπατε ότι βασικός στόχος είναι η δίωξη και η κατάσχεση των παράνομων εσόδων. Αυτό στη Μάλτα δεν συμβαίνει. Γιατί η αστυνομία ελέγχεται από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό και απλά δεν κάνει αυτά τα οποία εσείς λέτε και θέλετε. και η επιχείρηση αυτή η οποία είχε έδρα στο Ντουμπάι και κυκλοφόρησαν από τις τράπεζες στην Μάλτα και είχε ε, φυσικά σχέση ε, και με τους υπουργούς που υπέγραψαν τη συμφωνία για το φυσικό αέριο με το Ατζερμπαϊτζάν. Όλα είναι ένας κύκλος, σε πάση περιπτώσει. Τι κάνετε λοιπόν για να εντοπίσετε και να διώξετε τους ιδιοκτήτες και τους ε, υπεύθυνους αυτών των συναλλαγών και να κατασχέσετε τα κέρδη τους. Γιατί εδώ το βασικό θέμα το οποίο απασχολεί είναι η ε, γνώση του πραγματικού ιδιοκτήτη των επιχειρήσεων. Ας ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση να... πω ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής αξιολόγησης εφαρμόστηκαν όλοι οι κανόνες. Συντάξαμε επίσης και μία έκθεση. Η έκθεση αυτή δεν ζητήθηκε από την KPMG, αλλά από μία άλλη διεθνή εταιρεία η οποία χρησιμοποιείται από πολλές ρυθμιστικές αρχές μεταξύ των οποίων και την αρχή της Μάλτα. Δεν μπορώ να σας δώσω το όνομα της εταιρείας αυτής, χρειάζεται να ζητήσω την άδειά τους. Η έκθεση αυτή λοιπόν της δέουσας ε, που είχε σχέση με τον έλεγχο της δέουσας επιμέλειας, αν είχε υπάρξει, δεν ήταν πλήρης. Και στην ουσία ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αυτής ανήκε ουσιαστικά σε μία δικαιοδοσία η οποία σε επίπεδο νομικό παρουσίαζε ορισμένους κινδύνους και δεν υπήρξαν όμως κάποια στοιχεία ενημέρωσης τα οποία να είναι ανησυχητικά σε ένα πρώτο επίπεδο. Τώρα σχετικά με το κλείσιμο του πιστοτικού ιδρύματος, εμείς αμέσως ξεκινήσαμε την δίωξη σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές με στόχο όχι την ίδια την τράπεζα αλλά τον ιδιοκτήτη. Σχετικά με τις συναλλαγές τις οποίες είχε κάνει ο κύριος Σάντ, πριν εγκατασταθεί η συγκεκριμένη τράπεζα στη Μάλτα. Εμείς όταν αποδείξαμε ότι ο κ. Σάλντι ήταν ο βασικός μέτοχος, ξεκινήσαμε μια διαδικασία, ε, μια υπηρεσία εξωτερική να αναλάβει τον έλεγχο της τράπεζας, να ελέγξουμε ότι τα κεφάλαια της τράπεζας δεν θα έφευγαν και θέλω να πω ότι ήδη πριν από την ε, εκκίνηση της ε, διοκτικής διαδικασίας είχαμε ξεκινήσει μέτρα προστασίας και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται. Νομίζω ότι θα ελέγξουμε τελικά σύντομα το σύνολο των ισχυρισμών σχετικά με το αν έχει υπάρξει ξέπλυμα χρήματος από την τράπεζα. Όπως είπα οι ανακρίσεις συνεχίζονται. Περιμένουμε τα αποτελέσματα του συνολικού αυτού ελέγχου. Η κατάσταση είναι υπό εξέλιξη και όταν έχουμε τα τελικά στοιχεία, ανάλογα με το επίπεδο των στοιχείων, θα περάσουμε στα επόμενα βήματα. Σύντομα παρακαλώ. Θα είμαι σύντομος λοιπόν. Σχετικά με τις διώξεις ε, και τις κατασχέσεις προφανώς είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Δεν είναι εθνικό το θέμα. Αναγνωρίζουμε ότι και σε εμά είναι θέμα, αλλά είναι θέμα και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Δεύτερον, ε, σχετικά με την ανάλυση της συγκεκριμένης περίπτωση, εγώ δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες και ονόματα, αλλά θα ήθελα να σας ε, επιβεβαιώσω ότι αυτή στιγμή ε, ε, εμείς υποπτευθήκαμε ότι μπορεί να υπάρχει ξέπλυμα, στείλαμε μία αναφορά στις διοκτικές αρχές της χώρας μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που ήρθατε εδώ από τα εθνικά υποπτικά όργανα. Ε, θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση από την πλευρά των Ευρωβουλευτών ε, για να ακούσουμε την εμπειρογνωμοσύνη σας για πιο συστηματικά θέματα, όχι αναπερίπτωση, αλλά για καταστάσεις που αφορούν τα υποπτικά ζητήματα. Μήπως μπορείτε να προτείνετε κάτι πιο συστηματικό. Έχω λοιπόν τις εξή ερωτήσεις κυρίως στον κύριο Πούτνερς, αλλά ευχαρίστω αν και κάποιος άλλος μπορεί να απαντήσει. Καταρχάς χρειάζεται αυτή η λειτουργία ML σε, επίπεδο Τραπεζικής Ένωσης, δηλαδή είτε ΕΚΤ είτε Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, τουλάχιστον κάποιες μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης δεν συμφωνούν. Γι' αυτό θα είναι καλό βήμα αυτές οι χώρες που το επιθυμούν να το κάνουν. Έπειτα χρειαζόμαστε σε επίπεδο Eurozone κάποια ε, προειδοποιητικά μηνύματα που θα λένε ας πούμε ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλο ας πούμε, τομέα, πολύ μεγάλες τράπεζες ε, για αλλοδαπούς, ε, non-resident ε, και αυτό είναι κίνδυνος ή δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Τρίτο θέμα για τους ε, ψηφοφόρου μα, Πώ να εξηγήσουμε λοιπόν σε εκείνου, γιατί από καιρούς καιρών οι Αμερικανοί τιμωρούν κάποιες μεγάλες ε, τράπεζε, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη. Είναι ιδιαίτερε οι συνθήκε. Πώ μπορούμε λοιπόν να εξηγήσουμε, γιατί κάποιοι λένε ναι, η MBLV έχει κλείσει, αλλά κάποιοι μέτοχοι είναι κάποιε λουξεμβουργικέ τράπεζε. Και οι πελάτες που εξεκολουθούν να υπάρχουν στην ουσία ε, συνεχίζουν τη δουλειά τους με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι πελάτες είναι οι ίδιοι. Δηλαδή βασικά θέλουν να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν συναλλαγές σε δολάρια. Ε, μπορείτε να μας κάνετε κάποιες υποδείξεις για αυτό το θέμα. Κατά τη γνώμη σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε για την ε, ομοιόμορφη προσέγγιση για την υποπτία IML για την Ευρωπαϊκή Ένωση. να στηρίξουμε την, ε, ε, ε, το Εποπτικό Συμβούλιο και στο επίπεδο SSM, η κυρία Νούι είπε κάποια πράγματα στον τύπο σε σχέση με αυτό και προσωπική μου άποψη είναι ότι εγώ αυτό το στηρίζω τουλάχιστον για την Ευρωζώνη γιατί έχουμε ένα κοινό νόμισμα πράγμα το οποίο θα ε, πολλά χρήματα από το ελεκτικό σώμα AML. Το πρότυπο θα μπορούσε να είναι παρόμοιο όπως με το SSM, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή συγκεντρώνονται όλοι κάτω από την ε, αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όσον αφορά την Ευρωζώνη και το ξέπλυμα χρήματος, θα έλεγα ότι έχουμε δύο είδη μη ε, αλλοδαπών. Έχουμε μια ομάδα Έχουμε εκείνους ε, εκείνους που προέρχονται από, κυρίως από την Ρωσία, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που ε, αποτελούν μεγάλη απειλή τόσο για την εθνική μας ασφάλεια, όσο και για το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα που κινδυνεύει αλλά έχουμε και αλλοδαπούς από άλλες ε, χώρες της Ευρωζώνης, γιατί για τη Λετωνία έχουμε ε, Ουκρανού, ε, Ουκρανό, έναν Ουκρανό ή έναν Γερμανό. Και θα πρέπει να τραβήξουμε αυτή τη διαχωριστική γραμμή γνωρίζοντας την αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Δεν θα πρέπει να οικοδομήσουμε τείχους για να καταπολεμήσουμε αυτές τις καταστάσεις ε, ξεπλήματος χρήματος. Αυτή η διάκριση θα πρέπει να γίνει, αλλά να μείνει η ευρωπαϊκή μας αγορά ενοποιημένη και οι σχέσεις ε, όσον αφορά τους ε, αλλοδαπούς της Ευρωζώνης η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι τελείως διαφορετική από αυτήν που επιφυλάσσεται στους αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης. Τώρα, ε, χώρες εντός και εκτός Ένωσης, όπου όμως έχουν πολύ στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι ε, εάν ρευστοποιηθεί θα κλείσει η BLV. Δεν σημαίνει πως τα χρήματα θα πάνε σε κάποιες ε, χώρες του τρίτου κόσμου. Κατόλου. Η εντύπωσή μου είναι ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε πίσω στη Ρωσία. Και θα βρούνε το δρόμο τους ε, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι αυτό σημαίνει ενοποιημένη προσέγγιση, γιατί η τράπεζα στην ε, Λετωνία δεν σημαίνει ε, ε, σημαίνει ότι μπορεί να κλείνει οποιαδήποτε τράπεζα επειδή έχει γέφυρες με κάποια καθεστώτα και να υπάρχουν κάποιες τράπεζες αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα λες και δεν έγινε τίποτα. Είχαμε ορισμένε περιπτώσει τώρα με χρήματα από τη Βόρεια Κορέα. Δεν υπήρξε άμεση ε, ε, παραβίαση των ε, κυρώσεων ε, σε, για οποιαδήποτε τράπεζα της ε, Λετωνίας. Ε, ωστόσο, είδαμε ότι επειδή το πήραμε πολύ σοβαρά υπόψη και εξετάσαμε την κατάσταση, υπήρχαν έμεσες παραβιάσεις της, των κυρώσεων. Από όσο γνωρίζω όμως η Λετωνία ήταν η μόνη χώρα που έκανε κάτι τέτοιο. το ερώτημά μου είναι, ήρθε κατευθείαν στη Λετωνία ή πήγε αλλού πρώτα. Τα πήγαν αλλού πρώτα αυτά τα χρήματα γιατί τα χρήματα πέρασαν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και έφυγαν και από διάφορες δικαιοδοσίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και καμία άλλη δικαιοδοσία πουθενά δεν προέβη σε δράσεις κατά των τραπεζών που ήταν αναμεμειγμένες σε αυτή την υπόθεση. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Ε, για το υποτιθέμενο ε, ισότιμο πεδίο που ε, το λέμε και το ξαναλέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει αυτός ο ορισμός να πάρει σάρκα και οστά στην πραγματική ζωή. Ο κ. Στόρβαλτ. Ευχαριστώ. Λυπάμαι τελειώνει ο χρόνος, ε, μπορεί να επανέλθουμε στην γενικότερη ερώτηση εποπτείας ε, κάποια, στο θέμα της εποπτείας κάποια στιγμή αργότερα. Ο κύριος Τόρβαλς, ευχαριστώ πολύ. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα στοιχεία για τη Μάλτα. Και νομίζω ότι είπατε ότι δεν έχετε αρκετές ε, χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Ε, και μια ηρωνική, σαρκαστική απάντηση θα ήταν ε, ε, δεν αρκεί λίγη ευφυΐα. Εάν μια τράπεζα ονομάζεται Πιλάτος, ας, ας διαβάσει κανείς τη βίβλο ότι ένιψε τα σχήρας του. Όταν η Μάλτα ε, είχε την Προεδρία του Συμβουλίου, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για, την, για, για το ξέπλυμα χρήματος ε, και η Μάλτα πάντα πρόβαλε ε, εμπόδια όταν θέλαμε να εντοπίσουμε τους πραγματικούς δικαιούχους. Το 2015 το 30% των ε, νέων υπηκών της ε, Μάλτας ε, ήταν Ρώσοι, το 8% από το Ηνωμένο Βασίλειο και 4% από την Ουκρανία. Η οργάνωση της εταιρείας που οργάνωσε αυτό το καθεστώς θεωρήσεων Είναι γνωστό ότι κάναν το ίδιο για την Αντίγουα, την σε την Κύπρο, τη Γρανάδα, τη Μάλτα, Σέιν ε, Κίτς και, Saint... και Αγία Λουκία. Είναι όλες χώρες ε, που εμπλέκονται στα έγγραφα του Παναμά και των φορολογικών παραδείσων. Ακόμα δηλαδή και χωρίς ε, χρηματοοικονομικές πληροφορίες, με λίγη απλή ευφυΐα, θα έπρεπε να γνωρίζει κανείς ότι κάτι τρέχει. Και δεν είναι μόνο δικό σας πρόβλημα. Λέτε είναι ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα. Αλλά το δικό μου πρόβλημα είναι, είναι μαλτέσκο, το πρόβλημα μήπως είναι πανευρωπαϊκό. Σε ευχαριστώ, Νίλς. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Να συνεχίσω κι εγώ λίγο χιουμοριστικά. Εγώ από ό,τι γνωρίζω η τράπεζα λεγόταν Πιλάτος, όχι λόγω του, της βίβλου, αλλά λόγω του βουνού στην ε, Ελβετία. yes. Ε, the, the ε, member spoke. Ναι, ο, ο κύριος Ευρωβουλευτής Ε, μίλησε για τα εμπόδια που έθεσε η Μάλτα στη συζήτηση αυτή κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας της ε, όσον αφορά τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων. Εγώ διαφωνώ με τη θέση αυτή. Πιστεύω ότι... Πιστεύω ότι η Μάλτα ως Προεδρία έπρεπε να αντικατοπτρίζει τη θέση του Συμβουλίου. Είχαμε υποβάλει μια σειρά επικοδομητικών προτάσεων για το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι προσεγγίσαμε το στόχο μας, αλλά εκκρεμούν ακόμη κάποια ζητήματα και απαιτείται, απαιτούνταν περισσότεροι μήνες για να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι δυσκολεύαμε την κατάσταση. Ή ότι κολλησιεργούσαμε, θέλαμε μία καλή οδηγία, νομικά καλά στηριχμένη και λειτουργική στην πράξη. ενεργήσαμε με βάση τη θέση των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Όσον αφορά το IIP, δεν έχουμε καμία σχέση με το πώς διαμορφώθηκε και το πώς λειτουργεί και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τραπεζών όσον αφορά την νομοποίηση παράνομων εσόδων, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα κεφάλαια που εθνικοποιούνται με το σύστημα IIP, περνούν ε, τους σχετικούς ελέγχους που επιβάλλουν οι κανόνες. Εάν κάποιος ε, αγοράσει ιδιοκτησία στη Μάλτα, θα πρέπει να συνομιλήσει με εθνικές αρχές που επίσης θα πρέπει να κάνουν σχετικούς ελέγχους. Θα πρέπει επίσης ε, να έχουν επαφέ με συμβολιογράφου, που επίσης έχουν κάποιες υποχρεώσει. Περνούν λοιπόν από διάφορους ελέγχους. οι επενδύσεις των ανθρώπων αυτών που αποκτούν τελικά την μαλτέζικη υπηκότητα. Όσον αφορά τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας, Νομίζω ότι ακολουθούνται οι κανόνες, αλλά δεν μπορώ εγώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό, ούτε σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις. Πολύ σύντομα για το θέμα των χρυσών θεωρήσεων. Τι να σας πω για τις ε, χρυσές θεωρήσεις. Αυτή είναι η διαδικασία που περνάει κανείς για να ε, λάβει θεώρηση η υπηκότητα. Πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές για τα ζητήματα αυτά. Είμαστε ε, η εποπτική αρχή, δεν είμαι όμως η αρμόδια αρχή. Ε, ο κύριος Σατόραλτς, εγώ ρωτάω εάν είναι μαλτέζικο πρόβλημα ή αν είναι πρόβλημα της Ευρώπης όλης. Ε, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό αν έχουμε χρόνο στη διαδικασία Catch the Eyes. Παρακαλώ τους ε, ομιλητές ε, να τηρούν το χρόνο τους. Ε, Μόλις Σκοτ Κέιτο από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την Τράπεζα Πιλάτους ε, και ε, πρόσεξα τα γελάκια στην ε, αίθουσα ε, όταν, ε, δεν, όταν αρνηθήκατε να απαντήσετε ποιος έχει γράψει την έκθεση. Είναι δημοσιευμένη, νομίζω μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος την έγραψε. Όσον αφορά τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας, δώσατε στις 3 Ιανουαρίου του 2014 άδεια σε πρόσωπο για για τον οποίο ήδη είχαν ξεκινήσει ε, οι έρευνες και ε, είχε κατηγορηθεί ε, με έξι κατηγορίες για παραβίαση των κανόνων της των Ηνωμένων Πολιτειών για την νομοποίηση παράνομων εσόδων. Αλλά κάτι πάει στραβά εδώ. Πώς είναι δυνατόν να δίνεται υπηκότητα σε κάποιον που ήταν ήδη υποπτώσει για νομοποίηση παράνομων εσόδων. Σίγουρα κάτι έχει πάει στραβά. Και τέλος, ε, όσον αφορά τις ε, σχέσεις ανάμεσα σε και τράπεζες ε, και πολιτικά εκτεθμένους ανθρώπους από το Αζερβαϊτζάν, βλέπουμε ότι υπήρχαν επαφές με την οικογένεια της ηγεσία του Αζερβαϊτζάν και με επαφές με τη Γεωργία, το Μοντενέγρο, το Μαυροβούνιο και άλλα. Τι θα κάνετε στο μέλλον για να αποτρέψετε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Ίσως να μην ήμουν αρκετά σαφής. Η ανεξάρτητη έκθεση που ανατέθηκε κατά τη ε, διάρκεια της διαδικασίας για ε, την αδειοδότηση δεν ζητήθηκε από την KPMG, ζητήθηκε από διεθνή εταιρεία αλλά ε, ε, δεσμευόμαστε από τη σύμβαση να μην αποκαλύψουμε το όνομα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, για λόγους εμπιστευτικότητας ε, και συμβατικούς λόγους. Δεν ήταν η KPMG, ούτε η Μολτίζ ήτανε. Πρόκειται για εταιρεία που παρέχει πληροφορίες σε διάφορους Ευρωπαίους νομοθέτες και κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένων συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και τη ε, αρμόδια αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήταν ικανοί να διενεργήσουν μια ανεξάρτητη έρευνα. Όσον αφορά το γιατί δόθηκε στον κύριο Σάρντα άδεια να ανοίξει τράπεζα στην Μάλτα ενώ εκκρεμούσαν εις βάρος του έρευνες στις ΗΠΑ. Ε, η απάντηση είναι πολύ απλή. Κανείς εκτός των Ηνωμένων, Κανείς εκτός Πολιτειών ε, γνώριζε ότι ε, εκκρεμούσαν έρευνες εις βάρος του. Και καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της τράπεζες, συνεχίστηκαν οι εργασίες ε, με εφαρμογή της αρχής ε, της δέουσας επιμέλειας, με εκθέσεις που μας υποβλήθηκαν, αλλά δεν ε, ήταν δυνατόν με τα στοιχεία αυτά να γνωρίζουμε αμέσως ότι εκκρεμούσε έρευνα στις ΗΠΑ και όταν ενημερωθήκαμε γι' αυτό οι πληροφορίες που μας έδωσαν ήταν πάρα πολύ ισχνές. Δεν ε, γνωρίζαμε λοιπόν το πλαίσιο, δεν γνωρίζαμε το αντικείμενο των ερευνών, διότι σαφώς ε, οι αρχές των ΗΠΑ και το FBI δεν ε, διαδίδουν πληροφορίες στην διεθνή κοινότητα σχετικά με τις έρευνες που εκκρεμούν. Όσον αφορά λοιπόν τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας, δεν υπήρχε κανένας τρόπος να γνωρίζουμε ότι το πρόσωπο αυτό ε, αποτελούσε στόχο ερευνών στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Αυτό ενδεχομένως ε, να μπορεί να βελτιωθεί. Και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι εύκολο να βελτιωθεί η κατάσταση, διότι οι αρχές επιβολής του νόμου, οι ε, ερευνητικές αρχές έχουν βάσιμους λόγους που δεν μπορούν να αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες. Αλλά το θέμα αυτό σίγουρα αποτελεί σημαντική πρόκληση. Μια πρόκληση που αντιμετωπίζαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα γνωρίζοντας ότι εκκρεμούν έρευνες ε, αλλά χωρίς να γνωρίζουμε το αντικείμενο και ε, ρωτούσαμε, ζητούσαμε πληροφορίες, αλλά δεν μας δίνανε. Δεν μπορούν οι αρχές να αντιδράσουν με βάση ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Πρέπει να αναλαμβάνει κανείς δράση σε ρυθμιστικό επίπεδο, όχι με βάση φήμες, αλλά με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά αν είχαμε πάει στον κύριο Ασάρδε και του είχαμε πει ε, εκρεμούν έρευνες εις βάρος σας ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, ή δεν μπορούμε να σας δώσουμε την άδεια επειδή εκρεμούν οι έρευνες αυτό θα είχε βλάψει την έρευνα. Συχνά λοιπόν βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση διότι ακούμε φήμες, ψήθυρους ε, τις οποίε αφενός δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επειδή είναι επιβεβαιότητες, αφετέρου μπορεί να προκαλέσουμε προβλήματα σε ε, έρευνες άλλη χώρα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να καλωσορίσω ομάδα συνδικαλιστών ε, από τα εργοστάσια της Volvo στην ε, Σουηδία, που είναι προσκεκλημένη του Όλε Λούντβιξεν εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για τη δουλειά μας και, θεωρούμε, και το θεωρούμε και ενθαρρυντικό σημάδι. representatives. Uh, well, uh, it's a little bit surprising you are not, in your written answers you have already given us, ο κύριος Κούλογλου, έχω κάποιες ερωτήσεις προς τους εκπροσώπους της ε, Μάλτας. Με τις απαντήσεις που μας δώσατε μέχρι τώρα, δεν μας δώσατε πληροφορίες αρκετά σε σχέση με τα πολιτικά εκτεθειμένα άτομα στις τράπεζες πλάτους. Όχι μόνο ονόματα, δεν μας είπατε, αλλά ούτε και ε, νούμερα. Σύμφωνα με την ε, Δάφνη Καρουάνα Γκαλήθια, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν αναμειγμένοι, όπως η σύζυγος του Πρωθυπουργού, ο, Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Τουρισμού και ο Αρχηγός Επιτελείου του Πρωθυπουργού. Και αυτές οι αποκαλύψεις δόθηκαν στην Δάφνη Γαρουάνα Γαλήθια από έναν από τη Μαρία Εφήμοβα που ήταν πληροφοριοδότης. Οι Μαλτιδέζικες αρχές ήθελαν εκείνη να εκδοθεί στη Μάλτα, είναι τώρα στην Ελλάδα και η Δάφνη Καρουάνα Γαλήθεια ε, δολοφονήθηκε. Ε, μετά από τις αποκαλύψεις της Δάφνης και την, ε, την δολοφονία της, αυξήσατε εσείς την εποπτική δραστηριότητα για την Τράπεζα Πελάτους ή όχι. Και αν την αυξήσατε και ερευνήσατε, Θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται. Αν όχι, γιατί όχι. Τι είστε, ανίκανοι ή συνένοχοι. Η κυρία Σικλούνα. Καταρχάς θέλω να τονίσω ότι μας δεσμεύει η εμπιστευτικότητα όσον αφορά τα ονόματα. Δεν θέλω όμως αυτό να εννοηθεί ως ε, άρνηση συνεργασίας, αλλά ναι, δεσμευόμαστε από την εμπιστευτικότητα. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ονόματα ε, των πολιτών. Όσον αφορά την εποπτεία, φυσικά και έχουμε πλήρες λεπτομέρειες όσον αφορά την τράπεζα. Και όσον αφορά την εποπτεία, όπως σας είπα, στην αρχική μου δήλωση, Εμείς ε, άμεσα αντιδικοπαίσαμε την εποπτική μας ε, δραστηριότητα. Ας πάω, κάνω μια αναδρομή. Αυτή η τράπεζα ήταν από στενή εποπτεία εξ αρχής. Ξεκίνησε μια αρχική πλήρης ε, επιθεώρηση το 2017 από την μονάδα τραπεζικής εποπτείας. Τότε εμείς ε, θέλαμε να διαπιστώσουμε αν πληρούνταν οι όροι για την λειτουργία αυτής της τράπεζας. Σύμφωνα με τη Συμφωνία Συνεργασίας έγινε σχετική έκθεση και προς το FAEU που το Μάρτιο του 2015 μάλιστα διεξήγαγε επιτόπου επιθεώρηση, έλεγχο. Η MFC συμμετείχε σε αυτόν τον έλεγχο. Τον Αύγουστο του 2016 έγινε νέο, νέος έλεγχος, εν τω μεταξύ, ναι, συγγνώμη, αλλά μετά μάλλον σύμφωνα με τα, μετά από τα άρθρα της κυρίας Γαρουάνα Γκαλήθια, αυξήσατε την υποπτική δραστηριότητα και αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η ερώτησή μου και δεν μου απαντάτε. Μάλιστα, σίγουρα βεβαίως αυξήσαμε την ε, ε, ε, εποπτική διαδικασία που όμως είχε ήδη ξεκινήσει. Μάλιστα προέβημε σε διάφορες πρωτοβουλίες. Αυξήσαμε την ανεξάρτη τους ανεξάρτητους ε, ελέγχους πληροφορίες. Συνεργαστήκαμε στενά με τη ΦΕΙΓΙΟΥ και με άλλους διεθνείς ρυθμιστές. Ε, κάναμε περισσότερες ερευνές τόπο ε, και επιτόπιες και όλοι ε, σε αυτές οδήγησαν στη συγκέντρωση πληροφοριών που οδήγησε στην ολοκληρωμένη και εις βάθος εξέταση της έρευνας, δηλαδή ανάλυση όλων των λογαριασμών και των συναλλαγών, όπως σας είπα ώστε να έχουμε πιο στεναρή αξιολόγηση για το κατά πόσο η τράπεζα όντω συμμετείχε σε δραστηριότητε ε, ξεπλήματο χρήματο. Ε, ε, αυτό συνεχίζεται ακόμα. Αυτή η έλεγχη για να είναι αρκετά ολοκληρωμένη. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν τα πορίσματα θίγουν πολιτικούς. Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας, λέει η κυρία Σικλούνα. Πρόεδρος, ε, ναι, είναι ε, καυτά τα θέματα, αλλά παρακαλώ, εάν θέλετε να διακόψετε τον ομιλητή, ε, παρακαλώ κάντε το, ε, ενημερώστε με πρώτα. Κύριε Κούλογλου, θέλετε να παραλάβετε την τελευταία σας ερώτηση. Μάλιστα, είπα Υπήρξε επιπλέον εποπτική δραστηριότητα λοιπόν μετά από τους ισχυρισμού της Δάφνης Καρουάνα και η κυρία Σικλούνα λέει πως έχουν κάποιες απαντήσεις. Η ερώτησή μου είναι εάν αυτές οι απαντήσεις αγγίζουν, φύγουν πολιτικούς της χώρας. Ε, όπως σας είπα, ε, ο έλεγχος ακόμα γίνεται, η έρευνα ακόμα συνεχίζεται. Δεν είμαστε σε θέση να αποκαλύψουμε τα αποτελέσματα. Όταν θα αναλύσουμε ολόκληρη όλα τα αποτελέσματα, θα σας ενημερώσουμε. Πότε ξεκίνησε και πότε θα τελειώσει. Μπορώ να δώσω κάποιες πιο ε, πολλές λεπτομέρειες με τους περιορισμούς που μου επιβάλλονται. Πρώτα απ' όλα η απόφαση για να διεξαχθεί πολύ λεπτομερής έλεγχος και εξολόγηση και ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων της τράπεζας ελήφθη μετά το περασμένο καλοκαίρι. Και η διαδικασία επίσης αποφασίστηκε να ξεκινήσει τρίτο μέρος, να, μάλλον να συμμετέχει τρίτο μέρος, μια ειδικευμένη εταιρεία ε, πλήρως ανεξάρτητη για να βοηθήσει τις αρχές της Μάλτας. Βεβαίως... Ε, χρειάστηκε να ακολουθηθεί ε, διαδικασία διαγωνισμού, προκήρυξης διαγωνισμού και επιτόπια ε, η εργασία ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Σημαίνει πλήρη και βαθιά αξιολόγηση και έλεγχο των δραστηριοτήτων της τράπεζας, ε, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης όλων των διαδικασιών ανάλυση και εξολόγηση όλων των λογαριασμών που είχαν ανοίξει από την τράπεζα και αυτούς που είχαν κλείσει όμως, ανάλυση όλων των συναλλαγών που έχουν γίνει μέσα από κάθε ε, λογαριασμό, εισερχόμενες και εξερχόμενες ροές ε, χρημάτων. Από ποιον σε ποιον. Η ανάλυση επίσης περιλαμβάνει πλήρη αντιγραφή όλων των στοιχείων της τράπεζα, των εγγράφων, των email, των φωνητικών ε, καταγραφών και όλα αυτά αναλύονται από ειδικέ ε, ομάδες για να ανακαλύψουμε αν υπάρχουν συναλλαγές ή αποδείξεις για ξέπλωμα χρήματο ή άλλων μορφής εκκλήματος που θα μπορούσαν να έχουν κοινή επαφή με την τράπεζα. Η διαδικασία λοιπόν αυτή γίνεται εδώ και αρκετό καιρό, οπότε καταλάβαμε χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αρχίσουμε να έχουμε αποτελέσματα, τα οποία είναι ενδεικτικά για το πώς και πού μπορούν να, να, να, να, βρεθούν οι αποδείξεις που χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε φυσικά να ενεργήσουμε μόνο με ισχυρισμούς ή με βάση τα όσα γράφονται στις εφημερίδες ή με βάση πληροφορίες που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Χρειαζόμαστε σκληρές, σκληρά στοιχεία αποδείξεις και αυτή η προσπάθεια, αυτό το στόχο έχει να βρει τα στοιχεία. Και μετά θα μπορέσουμε να προβούμε στις απαραίτητες ε, οριστικές αποφάσεις. Εδώ μεταξύ έχουμε ε, εξασφαλίσει ότι η τράπεζα αυτή δεν λειτουργεί πια Όλα τα χρήματα έχουν παγώσει. Κανείς δεν μπορεί να πάρει χρήματα από την τράπεζα, ούτε να λειτουργήσει την τράπεζα με κανέναν τρόπο. Ο κόσμος ε, που δικούσε την τράπεζα έχει απομακρυνθεί. Ο έλεγχο ε, γίνεται από άνθρωπο που εμείς έχουμε ορίσει. Είναι για, ε, πρόκειται για ένα συνταξιούχο Αμερικανό ρυθμιστή με πάρα πολλή εμπειρία και Καθώς υπάρχουν προκύπτουν πληροφορίες από αυτή την προσπάθεια αλλά και από την ε, ανάλυση τη δική μας που ολοκληρώνεται θα ληφθούν και αποφάσεις. Η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ σύντομα. Είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε, όλες, σε λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων συντόμως. Και επίσης αναγνωρίζουμε πως η τράπεζα μπορεί να έχει βρώμικο χρήμα και είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε και αυτά τα χρήματα, αν υπάρχουν. Δεν νομίζω πως πρέπει να βιαστούμε. Πρέπει να τα κάνουμε όλα με τη σειρά τους. Να έχουμε σωστές πληροφορίες, να έχουμε αποδείξεις και να προστατεύσουμε οποιαδήποτε χρήματα πρέπει να προστατευτούν. Και σε περίπτωση που υπάρξει επιβολή ε, δράση μάλλον από τις αστυνομικές δυνάμεις μετά από τις ερευνές μας. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Η FTD δεν βλέπω κανέναν. Η ΕΝΕΦ θέλει κανείς το λόγο. Όχι. ΕΛΚ τώρα. Η Ρομπέρτα Μετσόλα. Ευχαριστώ πολύ. Ως μόνη Μαλτέζα σε αυτή την αίθουσα ε, θέλω να πω κάτι σαφέ. Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει τέτοιου είδου προκλήσει που δεν έχουμε δει εδώ και δύο γενε. είναι σημαντικό ο κόσμο που κοιτά προς την μικροσκοπική μας χώρα να γνωρίζουν ότι οι δράσει των εγκληματιών, των διεφθαρμένων στο ψηλότερο επίπεδο τη κυβέρνηση, δεν αντιπροσωπεύει το λαό τη Μάλτα. δεν εκπροσωπεί τη χώρα μου και το λαό μου, ε, δεν είμαστε παράδεισος φορολογικό, ε, δεν είμαστε δίκαιοι. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η δυνατότητα να ανταποκριθούμε, όπως ακούσαμε μόλις, έχει μειωθεί και αυτό είναι το τίμημα της διαφθοράς και της έλλειψης πολιτικής δράσης. Σε συγκεκριμένα ερωτήματα προς την FIAU θα προσθέσω στα όσα ήδη τέθησαν ως ερωτήσεις, αλλά δεν απαντήθηκαν. Γιατί πιστεύετε πως η αστυνομία, και πρέπει αυτό να το απαντήσετε, δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η έρευνα ε, σχετικά με κυβερνητικούς τους ε, πολιτικούς όταν γνωρίζουμε πως οι υπουργοί έχουν ε, πει ψέματα για λογαριασμούς που έχουν σε τράπεζες όπως αυτές ε, που εσείς ρυθμίζετε. Όπως γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον 200.000 ευρώ, δολάρια μεταβιβάστηκαν στο ε, Ντουμπάι μάλιστα ε, από πράκτορες του νέου μας ε, ε, ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού, όταν ξέρουμε πως οι υπουργοί είχαν λογαριασμού σε τράπεζες όπως οι πελάτες. Και αυτά δεν είναι φήμες, είναι, απο, είναι αποδεδειγμένα. Επίσης γνωρίζουμε ότι το FIU έχει στείλει εκθέσεις στον αστυνομικό διοικητή. Ποτέ δεν διερωτηθήκατε γιατί δεν έγινε τίποτα με βάση αυτές τις εκθέσεις. Και στην NFSA για την τράπεζα Τράπεζα Γνωρίζουμε πέραν πάση αμφιβολίες ότι πρόκειται για μια, ένα μηχανισμό ξεπλήματο χρήματο. Ο πρόεδρος τώρα σαπίζει σε μια αμερικανική φυλακή και ε, γνωρίζουμε επίση ότι όταν μας λένε ότι έγιναν επιτόπιε έρευνες, από ό,τι ξέρουμε είναι από διάφορου λέει ότι η Πιλάτους ήξερε ότι θα γίνουν επιτόπιε έρευνε είχε ενημερωθεί όταν όλες οι, οι κάμερες ε, του κόσμου κοιτούσαν τον Άλλη Σάντερ. Και θέλω να θυμίσω σε όσους ε, το μας ακούν ότι ο Πρωθυπουργός μας Μουσκάτ μετά τη συζύγου του μετέβησαν στο γάμο, ήταν καλεσμένοι στο γάμο αυτού του κυρίου στη Φλωρεντία πριν από λίγα χρόνια. Λέτε ότι δράτε με συγκεκριμένα, ότι δεν μπορείτε μάλλον να ενεργήσετε μόνο με ισχυρισμούς, φήμες, με συγκεκριμένες ε, πληροφορίες. Όταν όμως στέλνετε έκθεση Τη της FIU στην αστυνομία. Αυτό δεν είναι κανένα ψήθυρο. Αυτό είναι ορλιαχτό μέσα σε μικρόφωνο, σε μεγάφωνο. Ε, λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουν εκτεθεί στο δημόσιο χώρο θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχετε ενεργήσει πριν να δολοφονηθεί η Καρουάνα Γαλήσια. Έχουν τώρα επιβεβαιωθεί από τα πρακτορία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξέρουμε ότι ο Αλισάντερ είναι αυτός ο οποίος είναι αναμειγμένος σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εσείς δεν έχετε κάνει ακόμη τίποτα. Ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια του σε εμά και θα ήθελα πάρα πολύ να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί και να ξανακερδίσουμε την καλή μας φήμη που αυτή η κυβέρνηση έριξε στα σκουπίδια. Φαρούτσα. Ευχαριστώ κύριε Μέτσολα. Σχετικά με τις δράσεις των διοκτικών αρχών δεν είμαι εδώ για να τις σχολιάσω. Δεν μπορώ να ομιλήσω εκ μέρους της αστυνομίας της Μάλτα. Εγώ μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της αρχής την οποία εκπροσωπώ του ΕΦΑΙΟ. Έχουμε εκθέσεις ε, προσβάσιμες στην ιστοσελίδα μας, ανοιχτές, δημόσιες, μπορείτε να δείτε τι δουλειά έχουμε κάνει και σε επίπεδο συμμόρφωσης και σε επίπεδο χρηματοπιστωτικής ανάλυσης. Έχουμε στατιστικές ε, συνεργασίες ε, με ξένες υπηρεσίες. Όλα αυτά υπάρχουν και νομίζω ότι σαν οργανισμός μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όπως προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση της χώρας μου. Λοιπόν τώρα για την αστυνομία της Μάλτα εγώ δεν είμαι σε θέση να προσθέσω κάτι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και την κυρία Μέτσολα για την παρουσίασή της. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να πει κανείς ότι το MFSA δεν έχει κάνει τίποτα. Ήδη έχουμε εξηγήσει και λεπτομερώς μάλιστα το τι ακριβώς κάνουμε. Έχουμε ήδη εξηγήσει το τι μέτρα έχουμε συγκεκριμένα πάρει έτσι ώστε η τράπεζα να μην λειτουργεί στην παρούσα φάση Έχουμε πάρει μέτρα έτσι ώστε να προστατεύσουμε κάποιες καταθέσεις οι οποίες μπορεί να είναι ε, βρώμικες, να μην αποσυρθούν. Made it very clear that Έχουμε λοιπόν διευκρινίσει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ως ρυθμιστική αρχή δεν μπορούμε να αναλαμβάνουμε δράση με τις πληροφορίες των εφημερίδων μόνο. Εμείς παραπέμπουμε στις εκθέσεις της FIU, της ρυθμιστικής αρχής, not reports ε, οι εκθέσεις οι οποίες ε, έχουν κυκλοφορήσει δεν ήταν εκθέσεις για τη συγκεκριμένη τράπεζα αλλά για συγκεκριμένες ε, οντότητες οι οποίες χρησιμοποίησαν κάποιους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το ύψος των ποσών στα οποία αναφέρουν οι εκθέσεις αυτές που πέρασαν από την τράπεζα αυτή δύο ποσά των 50.000 ευρώ λέγεται στη μία έκθεση, στην άλλη έκθεση 9.500. Φυσικά και τα λάβαμε υπόψη μας, φυσικά και οι πληροφορίες αυτές μας ε, ενδιαφέρουν, μας ανησυχούν. But that αλλά η πληροφορία αυτή καθεαυτή ε, είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να ε, λάβουμε υπόψη μας αλλά φυσικά καμία ρυθμιστική αρχή ε, δεν θα έκλεινε μια τράπεζα γιατί είχε υποψίες για δύο ποσά 50.000 που πέρασαν από την τράπεζα. Προφανώς υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, ε, τις γνωρίζουμε τις πληροφορίες αυτές, τις γνωρίζαμε μετά από τη διαδικασία αδειοδότησης. Ε, γνωρίζαμε ότι ήταν υπό εξέταση το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο, ο βασικός μέτοχος. Είχαμε στοιχεία λοιπόν και αυτά ήταν τα στοιχεία τα οποία είχαμε επαναλαμβάνω. Εμείς πήγαμε επανειλημμένα, επισκεφθήκαμε την έδρα της τράπεζας, ζητήσαμε από την τράπεζα να αναφέρεται σε καθημερινή βάση και τώρα έχουμε ξεκινήσει θα έλεγα μια ιατροδικαστική έρευνα των δραστηριοτήτων της τράπεζας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω λοιπόν όλους σας και την κυρία Μέτσολα ότι και σαν ρυθμιστική αρχή και σαν ελεγκτική αρχή έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην ουσία και να βρούμε την αλήθεια του τι πρέπει να γίνει. Φυσικά και δεν είμαστε τέλειοι εκ των υστέρων όλοι μπορούν να τα κάνουν καλύτερα. Εγώ ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα που το σημειώνω αυτό. Αλλά εγώ, όπως είπε και ο Διευθυντής Φαρούτζα, μιλώ μόνο εκ μέρους της ρυθμιστικής αρχής και εν μέρη εκ μέρους της εποπτικής αρχής, της ελεγκτικής αρχής. Εγώ δεν θα σχολιάσω το τι έχουν κάνει οι πολιτικοί ή το ότι δεν έχουν κάνει, το ίδιο και για την αστυνομία. Εμείς ήρθαμε εδώ αποδεχόμενοι την πρόσκλησή σας, θέλουμε να είμαστε ειλικρινοί, δεκτικοί, αλλά μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας για αυτά τα οποία έχουμε κάνει ή για αυτά που δεν έχουμε κάνει. Δελβό, τελευταία ομιλήτρια, σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ. Μετά από την γεμάτη πάθος παρέμβαση της Μαλτέζας συναδέλφου, θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον λαό της Μάλτα και να εκφράσω τη διαμαρτυρία μου και την απογοήτευσή μου προς την κυρία Σίκλουνα γιατί δεν μας έδωσε το όνομα του προσώπου ή της εταιρείας της επιχείρησης η οποία έχει κάνει τον έλεγχο. Ίσως αν μας δώσετε μία γραπτή απάντηση να είσαστε κάπως πιο αναλυτικοί. Μία ερώτηση τώρα στον κύριο Πουτνινς για την ABVL. Ξέρω ότι υπάρχει συνεργασία με τις Λουξεμβουργιανές αρχές. Θα ήθελα να μας σχολιάσει τη συνεργασία αυτή και να πω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, τελικά πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται μόνο αν υπάρξει μια καταγγελία από κάποιον στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση αυτή κύριε Πούτνιενς. Ίσως τα επίπεδα συνεργασίας ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές και την ευρωπαϊκή ρυθμιστική δεν είναι τα κατάλληλα. Μήπως υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Και έρχομαι εδώ και στην προηγούμενη ερώτηση. Πιστεύετε ότι μια ευρωπαϊκή τέτοιου είδους αρχή, ένα ευρωπαϊκό FIU θα ήταν η κατάλληλη απάντηση. Λοιπόν, από τους ομιλητές ποιος θα πάρει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Η καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων είναι παγκόσμιο πρόβλημα και θα πρέπει να ε, εφαρμόσουμε παρόμοιες λύσεις και σίγουρα ε, είμαστε υπέρ της κεντρικής εποπτείας. Επειδή είναι παγκόσμιο θέμα, η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας. Έχουμε επενδύσει πολλά στη συνεργασία μεταξύ αρμοδίων αρχών από το 2014 και μετά. Ως επόπτης πρέπει κανείς να επιδιώχει τη συνεργασία. Νομίζω λοιπόν ότι η κεντρική προσέγγιση είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Πουτνίν ήδη απάντησε ή θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Ναι, να πολύ λίγα λόγια. Ναι, νομίζω ότι η ενιαία προσέγγιση είναι απαραίτητη. Και ο οργανωμένος έλεγχος των θεμάτων αυτών είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ιδέα, πολύ καλή πρωτοβουλία και θα πρέπει να συζητηθεί πώς είναι τεχνικά και νομικά εφικτό κάτι τέτοιο. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για τη μοναδική λύση εάν θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους παράνομων εσόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη. όσον αφορά την ε, APLV. Το πρόβλημα που ε, το πρόβλημα είναι ότι η διάταξη που εφαρμόζεται είναι τόσο αυστηρή που δεν υπάρχει ε, δυνατότητα διαμεσολάβησης. Σε άλλες περιπτώσεις όμως κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατόν. Αυτό λοιπόν που σκοτώνει την τράπεζα δεν είναι η στάση του επόπτη, αλλά η αντίδραση των αγορών και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Η ABLV λοιπόν θα διαλυθεί παρά το γεγονός ότι είχε μπει σε πρόγραμμα της FCMC η τράπεζα αυτή. Αυτό είναι ένα απλό γεγονός. Όσον αφορά τη συνεργασία μας με το Λουξεμβούργο, νομίζω ότι ήταν καλή. Ιδιαίτερα λόγω του ότι συνεργαστόμαστε στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και έχουμε πάντα τη δυνατότητα εκεί να συζητάμε διάφορα θέματα που προκύπτουν. Τότε που ήταν ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα το θέμα αυτό, ε, είχαμε επανειλημμένες έκτακτες διασκέψεις. Ε, εξαιρετική η συνεργασία μας λοιπόν με το Λουξεμβούργο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Σικλώνα. Εκτιμούμε αυτό που υπόθηκε σχετικά με την εταιρεία πληροφοριών που χρησιμοποίησαμε και θα υιοθετήσουμε την πρόταση του τελευταίου ομιλητή. Λυπούμε, δεν συγκράτησα το όνομα. Θα σας υποβάλουμε γραπτή απάντηση. Εάν συνενέσει η εταιρεία, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να σας αποκαλύψουμε το όνομά της. Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση σχετικά με τη συνεργασία. Στις παρατηρήσεις μας ε, υποβάλλουμε πρόταση για πιο ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στους επόπτες και ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές στις διάφορες δικαιοδοσίες. Υπάρχει περιθώριο για αυξημένη συνεργασία στον τομέα αυτών, κάτι που θα ε, κάνει πιο ορατές τις ρυθμιστικές αρχές και θα τους δώσει επίσης τη δυνατότητα να ενεργούν πιο ε, προορατικά. Και ναι, είμαστε εκεί πέρα ενό κεντρικού φορέα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι όλοι είναι υπέρ ενό κεντρικού συστήματος. Τρία ονόματα έχουμε με τη διαδικασία ΚΑΡΣΤΙΑΕ. Τον κύριο Καρίντς, την κυρία Ανακομές και την κυρία Ευαζολή. Θα ήθελα να τους παρακαλέσω να θέσουν πολύ σύντομες ερωτήσεις ε, και θα ακούσουμε πρώτα όλε τι ερωτήσεις και κατόπιν τι απαντήσεις. Ο κύριο Κάρινή, παρακαλώ. Ε, μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Νιώθω σαν να ξαναπρέθηκα εδώ. Είχαμε ε, οχτώ σκέψεις με την ε, Μαλτέζικη Προεδρία, με, ε, οχτώ ε, ε διαλόγους. δεν προχωρήσαμε όμως, μόλις με την επόμενη Προεδρία, την Εστονική Προεδρία προχωρήσαμε. Πώς λοιπόν συνέβη αυτό και να επανέλθω στην ε, Λετωνία. Κύριε Πούτνιν, αν κατάλαβα σωστά, λέτε ότι η APLV κατέρευσε λόγω της αντίδρασης των αγορών. Αυτό είναι λογικό. Ε, κλασική τράπεζα 600... Ε, ε, μια συνηθισμένη τράπεζα και ξαφνικά μαζική ανάληψη 600 εκατομμύριων. εκατομμυρίων. Ε, αυτό λογικό είναι. Αλλά ε, υπήρχε η ανακοίνωση της Φίνσεν ε, της Αμερικανικής ε, Αρχής. Ήταν σωστή, είχε δίκιο η Φίνσεν, το γιατί κατέρευσε η τράπεζα είναι δευτερευούσης σημασίας. Αλλά ε, ποιος ασχολιόταν με το θέμα του ξεπλήματος χρημάτων. Είχατε ασχοληθεί εσείς ή είχε δίκιο η Φίνσεν ότι δεν γινόταν τίποτα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε πρώτα ως ερωτήσεις η Άννα Καταρχάς ε, θα ήθελα να πω ότι θα στείλουμε στις ε, Μαλτέζικες Αρχές ερωτήσεις για να μας διευκρινίσετε τι μπορείτε να πείτε για το Black 17 ε, που ήταν δομή που υποτίθεται ότι ε, έπαιρνε χρήματα από διάφορους ε, που ε, νομοποιούσαν παράνομα έσοδα. Επίσης, φαίνεται ότι υπόθηκαν ψέματα στην Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Τι κάνετε για το θέμα αυτό και ε, οι πληρωμές από τη Βενεζουέλα στον κύριο Άλλη Σάντρ φαίνεται ότι περνούσαν από τις πορτογαλικές τράπεζες. Θα σας υποβάλω λοιπόν συγκεκριμένε ερωτήσεις και ελπίζω να μου απαντήσετε και εσείς γραπτός. Η ερώτηση μου τώρα είναι, αφού εστάλησαν οι εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τραπεζική Αρχή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι... Ε, αντίδραση είχατε εσείς ε, όσον αφορά τις αρμοδιότητές σας στον τομέα της νομοποίησης παρανομών εσόδων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζωλή. Έχω μια πολύ σύντομη ερώτηση για τον κύριο Φαρούτζια που είναι επικεφαλής ε, της ε, Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Θα ήθελα να γνωρίζω τι ενέργειες κάνατε όταν ε, είδατε ε, πολιτικούς με υψηλές θέσεις ε, να πηγαίνουν στο γάμο του προσώπου αυτού και Και εφόσον οι ιδιοκτικές αρχές δεν έδωσαν καμία συνέχεια στο θέμα, τι κάνατε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πούτνινς να απαντήσει τον κύριο Κάριν. Σας ευχαριστώ πολύ. η παρατήρησή μου είναι η εξής. Ε, η τράπεζα αυτή περνούσε από την ε, διαδικασία εξυγίανσης ε, και γιατί αποφάσισαν οι αρχές των ΗΠΑ να εκδώσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσουν οι εκπρόσωποι της Φίνσεν. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής, ότι το έγγραφο αυτό ποτέ δεν είχε στόχο να σκοτώσει την τράπεζα. Αν διαβάσετε τη δήλωση της Φίνσεν, είναι σαφές ότι προσπαθεί να προστατεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ και να αποκλείσει την ε, τράπεζα από την ε, περιοχή της. Αλλά η Φίνσεν αξιολόγησε τον κίνδυνο και αξιολογεί τη δυνατότητα να επιβιώσει η τράπεζα εκτός της ζώνης ε, του δολαρίου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν είχαν σκοπό να καταρρεύσει όλη η τράπεζα. Παρόμοια θέση είχαμε και εμείς και δεν είχαμε καμία αντίρρηση σε αυτά που έκανε η Φίνσεν. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να εξηγιάνουμε την τράπεζα. Η τράπεζα ήταν πρόθυμη να ε, συνεργαστεί και θα πρέπει να συμμορφωθεί. Και θα πρέπει να καταλάβουμε και το εξή, ότι υπάρχουν αρκετά σημαντικέ διαφορέ ανάμεσα στα νομικά συστήματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπη και ιδιαίτερα με τη Λετωνία. Η Φίνσεν λοιπόν λέει ότι η τράπεζα παραβίαζε το καθεστώς ε, των ε, κυρώσεων κατά της ε, Κορέας. Στις... Στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιος θα έπρεπε να διαπιστώσει ότι αυτό ήταν γεγονός. Το σύστημα στις Ηνωμένε Πολιτείες είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό της Ευρώπης. Κατά την ε, λήψη των ε, αποφάσεών μας, λοιπόν, εμείς ε, πρέπει να συμμορφωνόμαστε με το εθνικό μας δίκαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Σικλούνα. Θα, απαντήσω στην ερώτηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ε, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, είχαμε αρκετέ επαφές τον τελευταίο χρόνο για την υπόθεση αυτή. Είχαμε διάφορες ανταλλαγές πληροφοριών, συναντήσεις, τηλεφωνήματα και συζητήσεις πάνω στην υπόθεση αυτή. Έχουμε συνεχιζόμενες επαφές όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Γνωρίζετε ότι η αρχή ξεκίνησε μια προκατακτική έρευνα και είχαμε συζητήσεις και πλήρη συνεργασία μαζί τους. Η διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω, συνεχίζεται. Και σας διαβεβαιώ ότι θα υιοθετήσουμε οποιαδήποτε σύσταση της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής στο τέλος της έρευνας αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σπαρούτζη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ε, καλέσω την κυρία Γκόμες ε, να μας στείλει ε, ερωτήσεις στις οποίες ευχαριστώ θα απαντήσουμε. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών που ε, δέχτηκε την πρόσκλησή σας να έρθουμε εδώ να μιλήσουμε. Ε, θα καταλαβαίνετε όμως ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε συγκεκριμένες υποθέσεις λόγω εμπιστευτικότητας ε, και για να μην στρεβλώσουμε συνεχιζόμενες έρευνες. Θα κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά ε, την αστυνομία της Μάλτας, ε, στείλαμε εμείς στοιχεία στην αστυνομία. Κατόπιν η αστυνομία πρέπει να κάνει περαιτέρω έρευνες, ε, να διαβιβάσει, να μετατρέψει τις πληροφορίες σε αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν μπορούν να παρουσιάσουν στα δικαστήρια, πρέπει να βρουν λοιπόν αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια. Και αυτό απαιτεί αρκετό χρόνο, αυτό άλλωστε το ανέφερα στην ε, αρχική μου ομιλία. Και η αστυνομία πρέπει από, εκεί και πέρα να αναλάβει εκείνη την υπόθεση. Δεν μπορώ να σχολιάσω συγκεκριμένες υποθέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φαρούτζη. Ευχαριστώ όλους. Μία ακόμη ερώτηση για τους τριμερείς διαλόγους. Ε, θα παρακαλώ τον να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Σύντομα θα απαντήσω στην παρατήρηση του κυρίου Κάριν σε σχετικά με τα επιτεύγματα της Μαλτέζικης Προεδρίας και το θέμα ε, της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομοποίησης παρανομών εσόδων. Νομίζω ότι η Μαλτέζικη Προεδρία είχε επιτυχία όσον αφορά την πρόθεση της πρότασης για τον πραγματικό δικαιούχο εταιριών. και ακολουθήσαμε και τις ε, συμβουλές ε, της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Σε τεχνικό επίπεδο η Μαλτέζικη Προεδρία ολοκλήρωσε ε, σχεδόν το 60% του κειμένου συμπεριλάβαμε διατυπώσεις για την συνεργασία μεταξύ μονάδων χρηματοπιστωτικών πληροφοριών, για περισσότερο εις βάθος συνεργασία ανάμεσα στους επόπτες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι άδικο να λέτε ότι η Μαλτέζικη Προεδρία με τους περιορισμένους πόρους που είχαμε στην δυνατότητά μας δεν πετύχαμε τίποτα ε, στο θέμα της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κανείς άλλος να προσθέσει κάτι. Όχι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που ήρθαν εδώ. Και ε, όπως υπόθηκε μπορούν να, να υποβληθούν περαιτέρω ερωτήσεις γραπτός. Θα ήθελα να πω ότι και άλλη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών ε, αποδέχτηκε την πρότασή μας, αλλά είχε σήμερα άλλη συνάντηση με την Μάνιβα και γι' αυτό δεν μπορούσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Πάντως ε, θα κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά πάλι τη συζήτηση.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 Καλώς λοιπόν να ξεκινήσουμε το δεύτερο πάνελ. Όσοι μπαίνουν ή βγαίνουν αυτή τη στιγμή, παρακαλώ να το κάνουν γρήγορα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ε, το δεύτερο πάνελ για τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει τους σωστούς ελέγχους έτσι ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Ο κύριος Χάμπεν, υπεύθυνο για τις τραπεζικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, ο κύριος Μάριο Γκράντε, μέλος του SRB, ο κύριος Ρομπέρτο Γκουένα, υπεύθυνο νομικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ακούσουμε τρεις παρεμβάσεις από πλευράς τους. Και ο κάθε ομιλητής έχει στη διάθεσή του 7 λεπτά για να κάνει την εισαγωγή του. Technology. Thank you Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε στη σημαντική αυτή ακρόαση για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ε, για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και να ολοκληρώσω με κάποιες σκέψεις για το μέλλον. Νομίζω ότι θα γνωρίζετε όλοι την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και το ρόλο μας. Έχουμε πολλά καθήκοντα. Ένα από αυτά είναι να φροντίσουμε για την σωστή και συνεπή εφαρμογή της οδηγίας ε, κατά της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Να σας πω όμως κάποια πράγματα για το τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Ε, έχουμε κάποιες αρμοδιότητες, ε, κάποιες από αυτές είναι αρκετά ε, περιορισμένης λειτουργίες όπως είναι η δυνατότητα να επέμπουμε σε περιπτώσεις επίγουσες, αλλά ασχολούμαστε και με την ανάπτυξη προτύπων, με την κατάρτιση που είναι πολύ σημαντική για μας, αξιολογήσεις ομοτήμων και την διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών έχουμε ένα αρκετά ε, δυνατό εργαλείο που είναι η παραβίαση του ενωσιακού νόμου ε, που εξετάζει εάν εφαρμόζεται ο νόμος ή όχι και αν υπάρχει παραβίαση μπορούμε να υποβάλουμε συστάσεις ε, για να καλυφθεί αλλά δεν μπορούμε να φροντίσουμε για την για τις ελλείψεις κατά την εποπτεία και δεν είμαστε εμείς επόπτης ούτε επόπτης των εποπτών. Έχουμε κάνει πολλά όμως, νομίζω ότι οι οδηγίες 4 και 5 ήταν σημαντικά βήματα προόδου. η νομοποίηση παράνομων εσόδων είναι κάτι που αφορά πολλούς τομείς και πολλές χώρες και ξεπερνάει τα όρια του χρηματοοικονομικού τομέα η δουλειά που έχουμε κάνει. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα εντατική το, τους τελευταίους 18 μήνες και θα ήθελα επίσης την προσοχή σας σε κάποια θέματα. Έχουμε εκδώσει κατευθυντήρε γραμμέ για παράγοντε κινδύνου. Αυτό μπορεί να ακούγεται βαρετό, είναι όμω πάρα πολύ σημαντικό. 72 σελίδε με λεπτομέρειε σχετικά με τα θέματα που θα πρέπει να εξετάζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί όταν εξετάζουν τον κίνδυνο νομοποίηση παρανομών εσόδων και είναι και εργαλείο για τι αρμόδιε αρχέ για να αξιολογήσουν το πώ θα πάνε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Νομίζω ότι είναι πολύ πλούσια πηγή πληροφοριών και θα πρέπει να βοηθάει τους επόπτες να βρούνε ε, κοινό έδαφος. Επίσης, ε, έχουμε ε, κατευθυντήρες γραμμές εποπτείας για, που να βασίζεται σε κίνδυνο, που βοηθάει τους επόπτες να επιλέγουν πώς θα αξιολογούν τους κινδύνους. Βέβαια, μια προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο σημαίνει ότι δίνουμε προτεραιότητα σε ε, στις ε, περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος, ε, ενώ το αντίθετο είναι η περίπτωση όπου ελέγχονται όλα. Μια τέτοια προσέγγιση θα εφαρμοστεί φέτος και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα ποια θα είναι η αποτελεσματική προσέγγιση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Ένα άλλο θέμα που ξεκίνησε το 2016 ήταν η συνεργασία μεταξύ των εποπτών και νομίζω ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα πρόοδου. Η πέμπτη οδηγία για την κατά τη νομοποίησης παράνομων εσόδων αποτελεί σημαντικό εργαλείο και θα ε, εκδώσουμε ένα μνημόνιο κατανόησης για να βοηθήσουμε τους ε, συναδέρφους μας ε, στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ροή πληροφοριών σε όλη την ενιαία αγορά. Οι κατευθυντές γραμμές αυτές θα βασίζονται στην οδηγία, αποτελούν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι πιθανότατα και συνολική λύση για όλα. Ε, αυτά λοιπόν έχουμε κάνει, έχουμε δημιουργήσει το πλαίσιο και εγώ και οι συναδελφοί μου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τις αρμόδιες αρχές ε, κατά την εφαρμογή. Αναφέρθηκα ήδη στην κατάρτιση. 400 ανθρώπους ε, έχουμε για την ε, κατάρτιση πάνω στο νέο αυτό καθεστώς. Ε, είναι πολλοί άνθρωποι αυτοί στο δικό μας τομέα. Ε, έχουμε χρησιμοποιήσει λοιπόν το εργαλείο αυτό της ε, παραβίασης του ενωσιακού νόμου και ευχαριστούμε τους ευρωβουλευτές που έπεσαν την προσοχή μας στο θέμα αυτό. Το έχουμε κάνει αυτό στο παρελθόν με την Πορτογαλία, έχουμε υποβάλει σχετικές προτάσεις και αυτή τη στιγμή ε, κάνουμε προκαταρκτικές έρευνες για πιθανή παραβίαση του ενωσιακού νόμου στην Μάλτα και στη Λετωνία. Μόλις θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, πολύ ευχαρίστως θα σας εξηγήσουμε τα ευρήματά μας. Η ομάδα μου παρευρέθηκε νωρίτερα φέτος στη Μάλτα και ε, εργάστηκε πολύ εντατικά. Επίσης, ε, κονούμε στρατηγική που να ξεπερνάει τα όρια της αξιολόγησης ομοτήμων, ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε την εφαρμογή στις διάφορες χώρες. Χωρίς ισχυρή νομική βάση, αυτό γίνεται περισσότερο σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Εξετάζουμε λοιπόν τι κάνουν ε, και τους ε, δίνουμε συστάσεις για το πώς μπορούν να βελτιώσουν την εποπτεία τους στον τομέα της αντιμετώπισης της νομιμοποίησης παράνομων εισόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ευχαρίστω θα λάβουμε υπόψη μας προτάσεις ε, των Ευρωβουλευτών. Με αυτά τα βήματα πρόοδου λοιπόν βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, ε, πλησιάζουμε όμως τα όρια των ε, αρμοδιοτήτων μας και του δυναμικού μας. Ε, πόσους έχουμε που ασχολούνται με την νομιμοποίηση παράνομων εισόδων. Είχαμε έναν, τώρα έχουμε δύο. Έχουμε λοιπόν πολύ περιορισμένο δυναμικό. Βέβαια έχουμε και μια ευρύτερη ομάδα και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές. Φτάνουμε όμως τα όρια του δυναμικού μας και των αρμοδιοτήτων μας. Τρεις ε, τομείς ε, προτείνω να εξεταστούν ε, περαιτέρω εντός του ισχύοντος πλαισίου. Πολύ ωραία ιδέα του να έχουμε έναν επόπτη για την ομοιοποίηση παράνομων εσόδων, αλλά αυτό είναι ε, αυτό είναι θέμα εκτός του πλαισίου που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εντός του πλαισίου λοιπόν τι έχουμε, την ελάχιστη εναρμόνιση ε, που επιτρέπει τις ε, διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Θέλουμε σύγκληση λοιπόν διότι ε, οι σημαντικέ διαφορέ που υπάρχουν ε, εμποδίζουν ε, την σωστή αντιμετώπιση τη νομοποίηση παράνομων εσόδων. Επίσης, οι κανόνες για την αδειοδότηση, την ικανότητα των τραπεζών και την επιμέλεια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και την εθνική ερμηνεία. Σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές δεν μπορούν να αναλάβουν δράση κατά κάποιο ατόμο εκτός εάν υπάρχουν τελικά και οριστικά στοιχεία ε, ποινική ε, καταδίκηση. Νομίζω λοιπόν ότι και εδώ μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, να βελτιώσουμε την κατάσταση. και τέλος, εάν θέλουμε στην ε, Ευρώπη ανεξάρτητο έλεγχο της εφαρμογής από τις αρχές των κανόνων, νομίζω θα είναι χρήσιμο να έχουμε ε, τις ανεξάρτητες ε, αναθεωρήσεις εφόσον ε, έχουμε τις σχετικές αρμοδιότητες και το δυναμικό. Και επαναλαμβάνω, το δυναμικό. Επανέρχομαι λοιπόν στον ενιαίο επόπτη για την νομοποίηση παράνομων εσόδων. Ε, είναι σημαντικό όμω να αλλάξουμε και το πλαίσιο, διότι αν διατηρήσουμε το πλαίσιο που έχουμε και ε, φέρουμε και έναν ενιαίο επόπτη, τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν καλή συνεργασία και βέβαια ένας τέτοιο επόπτη θα χρειαστεί επίσης το απαραίτητο δυναμικό. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ σας ευχαριστώ, Κύριο Μάουρο Γκράντε από το νέο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτό το σημαντικό πάνελ. Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω την προοπτική υπό την οποία εξετάζει ο δικός μας οργανισμός την υπόθεση του ξεπλήματος χρήματος. Βασικός, βασική αποστολή είναι να εξασφαλίσουμε μια τακτική εξυγίανση μιας ε, τράπεζας που ε, καταραίει με ελάχιστο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία το θέμα της δομιμοποίησης παράνομων εσόδων δεν είναι πρωτογενές ε, καθήκον της αρχής εξυγίανσης. Η αρχή εξυγίανσης, ωστόσο, πρέπει να προσέχει και να μεριμνεί για όλες τις, εποπτή, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα υποθέσεις ξεπλήματος χρήματος στην εξυγίανση των ιδρυμάτων με τα οποία ασχολείται. Με αυτή την οπτική ε, εξετάζουμε το θέμα και πρέπει να σας προμολογήσω ότι μάθαμε πολλά από την υπόθεση BLV την οποία συζητήσατε στο προηγούμενο πάνελ. Πρώτο βασικό απόφθεγμα, δίδαγμα, είναι η ανάγκη εναρμόνισης ε, διεθνών, ε, διεθνώς του καθεστώτος ε, αφαιρεγγιότητας. Όχι μόνο για την ενιαία αγορά δηλαδή, είναι σημείο κλειδί γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει συσχέτιση από μία, ανάμεσα, μάλλον δεν υπάρχει συσχέτιση μιας τράπεζας που πτωχεύει, μπορεί να πτωχεύσει με την εξυγίανση σε τοπικό επίπεδο. Η, απο, η αναστολή Τη άδεια λειτουργία ε, είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Δηλαδή μπορεί να ρευστοποιηθεί μια τράπεζα με κατά μας, αλλά να συνεχίσει να δουλεύει σε εθνικό επίπεδο αυτή η τράπεζα. Αυτό πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε. Δεν υπάρχει αυτόματη συσχέτιση ανάμεσα στα δύο τώρα. Αναχέτηση του ξεπλήματο χρήματο. Αυτό που μάθαμε επίση από την εμπειρία είναι όταν σε μια περίπτωση μια τράπεζα επηρεάζεται από φήμε που σε αυτή την περίπτωση σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματο και αυτό δημιουργεί ε, προβλήματα ρευστότητα λόγω της αντίδραση αγορά, όπως είπαμε και πριν. Το θέμα είναι ότι επιδεινώνεται πάρα πολύ γρήγορα η κατάσταση τη Τράπεζα και φτάνει στο σημείο ε, κατάρρευσης πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση να λάβουμε σχετική απόφαση γρήγορα κι εμείς. Ε, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο μια κατάσταση όπου η τράπεζα πολύ γρήγορα ολισθαίνει προς μια τέτοια κατάσταση. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση της BLB, ε, μόνο 10 μέρες πέρασαν ανάμεσα στη στιγμή όπου μάθαμε τους κινδύνους ξεπλήματος χρήματος και την δήλωση της κατάρρευσης. Δέκα μέρες όλες και όλες. Αυτό είναι το θέμα, ε, ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί για την απόφαση εξυγίανση και να δράσουμε πολύ γρήγορα. Ποιοι είναι, ε, ποια είναι η πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρώτον, ε, να μιλήσουμε για την μοιρασιά ε, και την ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πολύ νωρί ε, του ισχυρισμού αυτού περί ξεπλήματος χρήματος για να μπορούμε να προετοιμαστούμε. Όμω το θέμα περιπλέκεται από το γεγονό ότι οι εθνικέ αρχές, ότι μάλλον οι αρχές που είναι υπεύθυνε για το ξέπλυμα χρήματο είναι σε εθνικό επίπεδο, ενώ εμεί είμαστε σε, σε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άρα εξαρτώμεθα από τις πληροφορίες που μας έρχονται από εκεί. Οτιδήποτε όμως επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφοριών θα μας βοηθήσει. Είμαστε νομίζω στην πέμπτη ε, αναθεώρηση της οδηγίας περί ε, ξεπλήματος χρήματος, οπότε οτιδήποτε βοηθά στην επιτάχυνση ανταλλαγή πληροφοριών και από νομοθετικής άποψης είναι πολύ θετικό. Το θέμα και η πρόκληση είναι η επιβολή αυτή της απόφασης ε, για μας. Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο κάθε τέτοια απόφαση. Το πρώτο σημείο λοιπόν σχετίζεται περισσότερο με το, τη στιγμή όπου ανακύπτει το πρόβλημα, αλλά εμείς ως αρχαία εξυγένσης πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για εξυγένση και στο πλαίσιο του προγραμματισμού του, της εξηγένσης είναι σημαντικό να μιλήσουμε με την, ε, τον επόπτη, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για το επιχειρησιακό μοντέλο. Ορισμένα ε, τέτοια μοντέλα, όπως γνωρίζουμε, είναι πιο ε, επιρρεπή σε τέτοια ζητήματα από άλλα. Εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά πρέπει να το γνωρίζουμε, ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε τις ε, δυνητικές περιπτώσεις, γιατί αν υπάρχει κίνδυνος τέτοιου ε, για, για φήμες, για καταγγελίες, θα είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί θα έχουμε πολύ μικρό χρόνο στη διάθεσή μας. Αυτό είναι μια κεντρική παρατήρηση. Αυτά λοιπόν κατά τη γνώμη μου περισσότερο έχουν να κάνουν με την λειτουργική πτυχή, επιχειρησιακή πτυχή, αλλά έχουν να ε, κάνουν και λίγο με ρυθμιστικά ζητήματα. Τώρα ευρύτερα για το ρυθμιστικό πλαίσιο, αν και δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό, εμείς υποστηρίζουμε αυτά που είπατε, ότι ε, την πιθανή εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου προς την κατεύθυνση περαιτέρω εναρμόνισης των ισχυωσών διατάξεων στον τομέα της ε, ε, του ξεπλήματος χρήματος, δηλαδή να κινηθούμε προς μια ευρωπαϊκή αρχή σε αυτό το τομέα, κατά την άποψή μας, είναι θετική. Θα έλεγα ως συμπέρασμα ότι εάν μας ρωτάτε ποιος, ποια μπορεί να είναι η συμβολή της εξυγίανσης στην ε, ανάσχεση του ξεπλήματος χρήματος, περισσότερο έχει να κάνει με την καλύτερη προετοιμασία σε περίπτωση που το θέμα ξεπλήματος χρήματος μεταφραστεί σε κίνδυνο από φημολογίες και καταλήξει σε μια κατάσταση όπου το να ολοκληρωθεί η εξηγήση μιας τράπεζας μπορεί να είναι πιο περίπλοκο. Να γνωρίζουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί όταν έρθει η στιγμή. Ενώ πώς θα μειώσουμε το κίνδυνο της ε, υλοποίησης αυτού του κινδύνου είναι περισσότερο τομέας ρύθμισης και εποπτείας εκεί. Ευχαριστώ για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και τις γραπτές απαντήσεις που στείλατε. Συγγνώμη. Θα δώσουμε και το λόγο στον κύριο Ρομπέρτο Ουγγένα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που έχω το λόγο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πριν περάσουμε στην ενίσχυση του πλαισίου καταπολέμησης του πλησίματος βρώμικου χρήματος, να αναφερθώ στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με τις προσπάθειες ε, για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Ε, Κάνοντας το αυτό νομίζω ότι οι απαντήσεις μου ίσως να είναι κάπως πιο χρήσιμες. Όσοι γνωρίσατε, ήσασταν μάλλον στην ακρόαση ε, ε του Προέδρου ε, της Εποπτικής Επιτροπής της Τράπεζας εδώ και ένα μήνα θα γνωρίζετε αυτά τα οποία θα πω. Η δημιουργία του ενιαίου ε, μηχανισμού εποπτείας έχει σαν στόχο όχι το να μεταφέρει αρμοδιότητες αλλά την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το άρθρο 127 παράγραφος 6 της Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν ε, η νομική βάση για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό περιλαμβάνει όρια και σε σχέση με την εμβέλεια των εποπτικών αποστολών τις οποίες μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και των ε, οντοτήτων που θα μπορούσαν να ελεγχθούν η εφαρμογή και η επιβολή ε, μέτρων ε, για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος, τα λεγόμενα AML, δεν είναι πλήρης αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όμως συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνε για το AML. Αυτή η κατανομή των αρμοδιοτήτων σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να είναι ικανή να μεταφέρει τα ευρήματα και τις ανησυχίες των εθνικών αρχών και στα πλαίσια της προληπτικής εποπτείας και στα πλαίσια της ενημέρωσης. Τώρα να σας πω πώς δουλεύει αυτή η κατανομή κατά κάποιο τρόπο και διάδοση των αποτελεσμάτων σύμφωνα ε, με την προσπάθεια την οποία κάνουμε σε ετήσια βάση, εξετάζουμε την ανάγκη για μέτρα στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα, λαμβάνουμε υπόψη και τους νομικούς κινδύνους και το κόστος το σχετικό με ποινικέ διώξεις, αλλά και θέματα φήμης, θέματα λειτουργίας, διακυβέρνησης και άλλες σχετικές πληροφορίες χωρίς τις πληροφορίες που παίρνουμε από τις εθνικές ελεγκτικές αρχές οι δυνατότητές μας είναι πολύ περιορισμένες. Στην περίπτωση απόσυρσης ή κατάργησης της τραπεζικής αδειοδότησης που γίνεται σε συνεργασία και με τον ενιαίο μηχανισμό με τις εθνικές αρχές, το γεγονός όμως ότι οι αρμοδιότητες έγκυνται σε εθνικό επίπεδο σημαίνει ότι η διαδικασία απόσυρσης της άδειας λειτουργίας ανήκει στις εθνικές αρχές και βασίζεται σε εθνικές ρυθμίσεις. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε ενήμεροι από τις αρχές αυτές για όλες τις αιτίες που οδηγούν στην απόσυρση της άδειας. Επί τη βάση των αξιολογήσεων που γίνονται από τις ε, αρμόδιες για το ξέπλυμα αρχές και στο εσωτερικό των αρμοδιοτήτων και του Εθνικού Νόμου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία αυτά. Να υπογραμμίσω ότι στα πλαίσια του εντοπισμού των κινδύνων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ε, ανεξάρτητα από τις εθνικές αρχές ε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι σαφές ότι τα περισσότερα εξαρτώνται από την προληπτική δράση των εθνικών αρχών και την ενημέρωσή τους προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η νομοθετική διαδικασία που θα οδηγήσει στην οδηγία AML5 θα βοηθήσει την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με το ξέπλυμα, δίδοντας μια πραγματική ισχυρή νομική βάση. Βέβαια απαιτείται μια πιο ευρωπαϊκή αντιμετώπιση στην καταπολέμηση του ξεπλήματος ρώμικου χρήματος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις ε, νομικές και εποπτικές δυνατότητες τις οποίες έχουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα και οι προληπτικοί επόπτες, η προληπτική εποπτεία που δεν είναι άμεσα αρμόδια για θέματα ξεπλήματος μπορούν να συμμετέχουν στις διεργασίες ως παρατηρητές. Οι συνάδελφοι τα εξήγησαν αυτά καλύτερα από μένα. Να υπογραμμίσω λοιπόν ότι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η δυνατότητά μας ως εποπτικού ελέγκτη έχει μεγάλη σημασία να έχουμε έγκαιρες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του βρώμικου χρήματος, επειδή δεν είμαστε άμεσα υπεύθυνοι, εξαρτώμεθα από την συνεργασία μας με τα εθνικά επίπεδα ελέγχου για να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε στην εποπτική μας δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Ένα λεπτό θα έχει ο κάθε ομιλητής και τρία λεπτά για την απάντηση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ήθελα να ελέγχετε το χρόνο τον οποίο έχετε στη διάθεσή σας, παρακαλώ. Να προσπαθήσετε να σεβαστείτε τον χρόνο τον διαθέσιμο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας σήμερα. Είναι σαφής η ποικιλομορφία όσον αφορά την συνεργασία και αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Πόσο μάλλον όταν βλέπουμε και τη συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Υπάρχουν κενά εδώ. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον συντονισμό, την εναρμόνιση, ώστε να έχουμε ε, αποτελεσματική εποπτεία για την αντιμετώπιση της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Άκουσα αυτά που είπε ο εκπρόσωπος του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Είναι ντροπή το ότι έχουμε ένα σύστημα στην Ευρώπη όπου η κεντρική αρχή να μην έχει τη δυνατότητα να επέμβει σε, περίπτωσεις, σε περιπτώσεις νομοποίησης παράνομων εσόδων. Και πολλά κράτη-μέρη δυσκολεύονται πολύ να κάνουν τη δουλειά σωστά. Μια ερώτηση ίσως προς τον κύριο Χάρπεν. Μήπως μπορείτε να μα πείτε ποια είναι τα πιο προβληματικά κράτη-μέλη στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Χάμπεν βλέπω ότι βγάζει ένα κατάλογο από το, από το χαρτοφύλακά του. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Στο ισχύον πλαίσιο, όσον αφορά την ε, ενίσχυση της εργασίας και των ε, ροών πληροφοριών, η πέμπτη οδηγία νομίζω ότι δεν θα τα ανατρέψει όλα, αλλά θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Και εμεί, ε, λοιπόν πέρα από το Μνημόνιο Κατανόηση, ε, έχουμε ξεκινήσει την εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στι αρμόδιε αρχέ. Και με τις κατευθυντήρε αυτές γραμμές και αν έχουμε τη δυνατότητα ε, να ε, ελέγξουμε την εφαρμογή των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών, τότε πιστεύω ότι θα δούμε ενισχυμένη συνεργασία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε εντατικά. Δηλαδή και την εκπόνηση των κατευθυντήριων γραμμών και τη συνεργασία με ε, αρμόδιες αρχές για να καταλάβουμε τα εμπόδια στην συνεργασία που αντιμετωπίζουν. Στις απαντήσεις για τα έγγραφα του Παναμά ε, ρωτήσαμε διάφορους τι ακριβώς κάνουν και πάνω από το μισό των εποπτών ε, είχαν ήδη αναλάβει επιπλέον βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος όσον αφορά τις χώρες που δεν συνεργάζονται. Όταν ε, ζητάω ε, ανάδραση, όταν ζητάω στοιχεία από τους επόπτες μας, ε, λαμβάνω απάντηση, αλλά μπορώ να σα διαβάσω τον κατάλογο αυτών από του οποίου είχαμε αρνητική απάντηση. Ο Γέπε ε, είναι πολύ σύντομα. Αναφέρατε ότι η πέμπτη οδηγία επιφέρει ασφάλεια δικαίου και ότι κάποια νέα στοιχεία θα βελτιώσουν τη συνεργασία. Νομίζω όμως ότι πάλι το θέμα είναι απόκειται στις αρμόδιες αρχές, ε, στις εθνικές αρχές διαβάζω τις απαντήσεις σας, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτά αρκούν για να αντιμετωπίσουμε ικανοποιητικά το θέμα της νομοποίησης παρανομών εσόδων. Να ρωτώσω λοιπόν τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Δεν θα ήταν καλύτερο να έχουμε κεντρική εποπτεία ε, όσον αφορά την νομοποίηση παράνομων εσόδων και τι ρόλο παίζει ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός στο θέμα αυτό. Παρακαλώ, θα ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντας κάτι που υπόθηκε πριν, ότι δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε την αξία της αναθεώρησης της οδηγίας. Έχει για μας δύο σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με πριν. Καταρχάς, σαφής νομική βάση για την ανταλλαγή δεδομένων. Αυτό μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά στο παρελθόν δεν είχαμε αυτή τη νομική βάση και συχνά αντιμετωπίζαμε δισταγμό, θα έλεγα, για την ανταλλαγή πληροφοριών λόγω της έλλειψης σαφού νομική βάσης. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ αρνητικό. Και το άλλο που ανέφερε και ο Πίρς πριν, ε, τα μνημόνια κατανόησης. Νομίζω ότι θα είμαστε σε καλύτερη θέση με αυτά, διότι θα έχουμε τη δέσμευση των ε, αρμοδίων αρχών ε, να μοιραστούν πληροφορίες μαζί μας. Ενώ τώρα βασιζόμαστε περισσότερο στην ίδια πρωτοβουλία, ενώ στο μέλλον θα έχουμε δεσμεύσεις στα μνημόνια για την ανταλλαγή πληροφοριών. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι αυτά είναι σημαντικά επιτεύγματα κατά τη γνώμη μας. Πώς να προχωρήσουμε από το κεμπρός. Καταρχάς, θα ήθελα να σας θυμίσω αυτό που είπα στην αρχή. Ε, μπορεί το SSM να παίξει σημαντικότερο ρόλο. Θα πρέπει να πω ότι η συνθήκη θέτει κάποια όρια. Ε, για παράδειγμα το άρθρο 127 παράγραφος 6 της συνθήκης. ε, μας παρουσιάσει μια δυσκολία την οποία θα πρέπει να ξεπεράσουμε ε, αν θέλουμε να έχουμε έναν κεντρικό επόπτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να είναι αρμόδιος για θέματα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. τίθεται και το θέμα αν μπορούμε να αναλάβουμε και άλλα καθήκοντα, διότι τα συγκεκριμένα καθήκοντα τα ε, θέτει η συνθήκη. Έχουμε λοιπόν κάποιους περιορισμούς. Πέρα από αυτό όμως, τίθεται το θέμα αν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τις ικανότητές μας ως ε, φορέας. Ε, υπάρχει επιφύλαξη στον τομέα αυτό, ήδη έχουμε πολλά ε, καθήκοντα, αλλά δεν υπάρχει επίσημη απάντηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω οριστική θέση. Ευχαριστώ πολύ, Ντάριος Ρωσάτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και έχω να ευχαριστήσω τους ε, προσκεκλημένους μας σήμερα το πρωί. Στην πρώτη συνεδρία που είχαμε το πρωί, συζητήσαμε τρεις υποθέσεις τριών τραπεζών σε τρία κρατημέλη. Όπου διαπιστώθηκαν υποθέσεις παράβασης ε, της ε, νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης παράνομων προσόδων της Ένωσης. Στις τρεις περιπτώσεις όμως ε, το κόδωνας κινδύνου ήχησε στη ΣΥΠΑ. Οι ευρωπαϊκές οι εθνικές αρχές δεν είχαν ενημερώσει. Μπορεί και μην, να μην τις ήξεραν καν, εν πάση περιπτώσει ενημέρωναν με καθυστέρηση. Ποιος είναι ο λόγος, πού οφείλεται για αυτή η παράξενη κατάσταση, δηλαδή το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών να έχει μια, ε, ένα ειδικό τμήμα ε, που ασχολείται με τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί, γιατί είναι πιο αποτελεσματική η νομοθεσία αμερικανική ή επειδή η, η δημοσιονομική εποπτεία χρηματοπιστωτική εποπτεία σε αυτές τις χώρες δεν είναι αρκετά αποτελεσματική, είναι εξαιρετικά επίοικης. Ή δεν είναι αρκετά ενήμερη. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Στην πρωινή συζήτηση ένας από τους ε, προσκεκλημένους από τη Μάλτα είπε ο, ισχυρίστηκε ότι είναι απολύτως αθώοι για την υπόθεση του Τράπεζα της Τράπεζας Πιλάτο, ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη οι εθνικέ αρχές. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι παράξενο, γιατί αν γνωρίζουμε ότι... Ε, υπάρχει το σύστημα παρακολούθησης ε, της καταπολέμησης των, των ε, των ε, δραστηριοτήτων ξεπλήματος χρήματος. Αυτό είναι ευθύνη των εθνικών αρχών. Αυτές έχουν την πλήρη ευθύνη για, την οικονομ... για τα θέματα αυτά. Εσείς μοιράζεστε την άποψή μου και ότι δεν υπήρξε αρκετή συνεργασία και ότι αν υπήρχε τέτοιες υποθέσεις όπως η υπόθεση της τράπεζας Πιλάτους δεν θα, δεν θα είχαν ε, συμβεί. Σας ευχαριστώ για τις σημαντικές ερωτήσεις σας σε σχέση με τα θέματα που έθεσαν οι Αμερικανικές αρχές. Είχαν τεθεί κάποια ερωτηματικά και στην Ευρώπη. Υπάρχουν ε, δύο υποερωτήσεις. Καταρχάς, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές και δεύτερον, αν ήμασταν πιο δραστήριοι ή αν θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο δραστήριοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς δεν έχουμε σαν υπηρεσία τα μέσα και τις αρμοδιότητες να κάνουμε ανακρίσεις εξ αρχής και απλά καλούμεθα να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα δεδομένα και τις διαθέσιμες πληροφορίες. Τώρα, για την συγκεκριμένη τράπεζα Πιλάτους είναι η ευθύνη στην Εθνική Αρχή Έχουμε κάποιες δυσκολίες σε επίπεδο συνεργασίας και αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις μορφές συνεργασίας. Δεν ξέρω αν οι προτινόμενες αλλαγές είναι επαρκείς έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Πάντως υπάρχει θέμα δικαιοδοσίας και καλό θα ήταν να ήταν ενιαία η αντιμετώπιση των και καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος στο σύνολο της Ένωσης. Ο κύριος Σουχένα. Δεν νομίζω ότι απλά είναι θέμα συνεργασίας. Έρχομαι από μια χώρα όπου πριν από την δημιουργία του ενιαίου μηχανισμού η αρμοδιότητα για το ξέπλυμα, για την αντιμετώπιση δεν ήταν μια αρμοδιότητα η οποία ανήκε αποκλειστικά στον, στο επίπεδο της εποπτικής προληπτικής αρχής. Δεν είναι η αρμόδια αρχή λοιπόν και θα πρέπει όμως οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται γενικότερα σε όλα τα επίπεδα όταν προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν τα πιστοτικά ιδρύματα να τις έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με τις χώρες τις οποίες αναφερθήκατε. Η συνεργασία με εμάς ως εποπτική προληπτικά αρχή έχει, θα έλεγα, λειτουργήσει στο εσωτερικό του συστήματος αρκετά ικανοποιητικά. Τώρα, οι τα καθυστερημένα ευρήματα και οι διαδικασίες οι οποίες ξεκίνησαν με κάποια υστέρηση χρονική στις διάφορες χώρες δεν είναι θέμα συνεργασίας, είναι θέμα αρχιτεκτονικής εποπτικής ε, στις ε, διάφορες χώρες. Πάντως, στις δύο περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε, η συνεργασία μας με τις αρμόδιες αρχές πήγε καλά. Θα μιλήσω ισπανικά. Τρεις ερωτήσεις. Είναι σαφές ότι πράγματι απαιτείται να αλλάξει η νομοθεσία έτσι ώστε να υπάρξει ε, μεγαλύτερη ε, δυνατότητα και μεγαλύτερες εξουσίες στις εποπτικές αρχές. Σε σχέση με την δυνατότητα η εποπτική αρχή να καλύψει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να, να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιστεύετε ότι το Brexit θα επηρεάσει αρνητικά το σύνολο της εποπτικής διαδικασίας, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε ίσως να εκμεταλλευτούμε την δυνατότητα να έχουμε από του χρόνου η εποπτική αρχή να καλύπτει 27 χώρες. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει κάποιος συσχετισμός ανάμεσα στους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους και το ξέπλυμα. Τι ελέγχους ναι. κάνει η Κεντρική Τράπεζα και ο Μηχανισμός Εποπτείας και η EBA για τις ε, Ευρωπαϊκές Τράπεζες οι οποίες έχουν θηγατρικές εταιρείες σε δικαιοδοσίες τις οποίες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι ανήκουν στον λεγόμενο μαύρο κατάλογο ή στον θεό κατάλογο, τον γκρίζο κατάλογο. Δηλαδή δικαιοδοσίες οι οποίες δεν συνεργάζονται ως πρέπει. Και μια τελευταία ερώτηση, Πρόεδρε. θα ήταν θετικό για την καταπολέμηση του ξεπλήματος να υπάρχει ένα ενιαίο ανώτατο όριο της χρήσης μεταλλικού χρήματος στα πλαίσια των πληρωμών, των λιανικών πληρωμών.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 ε, ξεκινήσω εγώ και μετά θα συμπληρώσουν οι συνάδελφοι. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, εάν υπάρχει δυνατότητα να διευρύνουμε το πεδίο του SSM σε ολόκληρο την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περισσότερο πολιτική φύση το ερώτημα κατά πόσο δηλαδή υπάρχει διάθεση σε πολιτικό επίπεδο να γίνει κάτι τέτοιο και αυτό απαιτεί από την νομική άποψη την τροποποίηση του κανονισμού SSM που πρόκειται για έναν κανονισμό που εγκρίνεται μέσω μιας πολύ ιδιαίτερη νομοθετική διαδικασία όπου χρειάζεται ομοφωνία σε επίπεδο ε, συμβουλίου. Οπότε θα έλεγα λοιπόν ότι είναι περισσότερο πολιτικής, ε, πολιτικό το ζήτημα. Εάν υπάρχει διάθεση δηλαδή να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση ή όχι. Σε σχέση τώρα με δικαιοδοσίες που να μην είναι συνεργάσιμη όσον, συνεργάσιμες όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για το στόχο της καταπολέμησης του ξεπλήματος ε, χρήματος. Ε, εμείς είμαστε η αρμόδια αρχή, ε, είμαστε οι εποπτές για το για τον ομάδα, για τον όμιλο και φυσικά προσέχουμε και τις περιπτώσεις ε, όπου πρέπει να υπάρχει πιο στενή παρακολούθηση. Αυτό που κάνουμε είναι ετήσια εποπτική έκθεση που κάνουμε για κάθε τράπεζα για, την οποία είμαστε υπεύθυνοι. Ε, δηλαδή, αναλύουμε πολλά στοιχεία, αλλά ανάμεσα στα στοιχεία ε, αυτό που προσέχουμε είναι το επιχειρηματικό μοντέλο, είναι ένα εξ αυτών, και ο Μάουρο το ανέφερε προηγουμένως, στις εισαγωγικές του παρατηρήσεις. Όταν δηλαδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μοντέλα ιδιαίτερα όπου ας πούμε έχουν ε, ε, θηγατρικές σε αυτές τις χώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προκύψουν ζητήματα ε, ξεπλήματος χρήματος τότε ακολουθούμε το σύστημα των, της βαθμολογίας. Όσο μεγαλύτερο εκτιμούμε τέτοιο κίνδυνο, τόσο μεγαλύτερο σκόρ έχει αυτή η τράπεζα. Και Ζητάμε συγκεκριμένες ε, απαιτήσεις ε, ρευστότητας ε, ή άλλου είδους μέτρα πετούμε για την λογοτράπεζα. Τώρα, η EPA, αν είναι καλά, ε, αν είναι στην κατάλληλη θέση και να εκτιμά τις ε, ε, διάφορες συναλλαγές, νομίζω πως αυτό αυτό έχει ήδη γίνει σε κάποιες χώρες, έχει ήδη εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες και θα ήταν ίσως καλό να εξετάσουμε παραδείγματα αυτών των χωρών για το κατά πόσο στην πράξη ήταν αποτελεσματικό αυτό ή όχι. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σχάβεν. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Όσον αφορά το αν το Brexit αποτελεί ευκαιρία για να λύσουμε το θέμα αυτό, νομίζω ότι τώρα είναι η χρονική στιγμή να το λύσουμε. Δεν νομίζω το να αφαιρέσουμε μία χώρα από την εξίσωση θα αλλάξει την κατάσταση. Για άλλους λόγους λοιπόν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Άλλωστε διαπιστώσαμε ότι είναι εκτενές το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν αφορά λοιπόν μόνο μία δικαιοδοσία, αλλά σίγουρα τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή όσον αφορά τις εγκαταστάσεις σε δικαιοδοσίες, αναφέρεστε σε δικαιοδοσίες της μαύρης λίστας της FATF, της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Υπάρχουν λοιπόν ε, κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται και ε, αν γίνεται ετησίως ε, ο κατάλληλος έλεγχος σε επίπεδο ομίλου, τότε νομίζω ότι θα είναι και αποτελεσματικά τα μέτρα για τις ε, εγκαταστάσεις. Γι' αυτό είναι περισσότερο θέμα εφαρμογής των κανόνων. Ε, το σχετικό πρότυπο ε, θα δημοσιευτεί σύντομα. Πάντως συνδέονται τα δύο αυτά θέματα μεταξύ τους, δηλαδή το θέμα του πώς μπορούμε να αποκτήσουμε δεδομένα των πελατών. Επίσης, Οι μεγάλες ε, συναλλαγές με μετρητά είναι ένας από τους παράγοντες κινδύνου που θα πρέπει να εξετάζουμε και πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι μπορεί να υπάρχουν ε, συνέπειες ε, απρόβλεπτες, μεγάλες Μεγάλοι οργανισμοί ε, βοήθεια, βοήθειας, για παράδειγμα, μας λένε ότι χρειάζονται μεγάλες συναλλαγές μεγάλου όγκου μετρητών για διάφορες δικαιοδοσίε σίγουρα, μάλλον είναι ο κατάλληλος τρόπος να προχωρήσουμε το να εξετάζουμε τις ε, μεγάλες ε, συναλλαγές πάντως. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ ο κύριος Σίλα από το ECR. Ναι, όχι, έκανα λάθο ο κύριο Κράντε. Ε, ναι, συγχωρήστε με, απλά για να μην μείνω τελείω εκτό τη συζήτηση, αν και αναγνωρίζω ότι οι περισσότερε ερωτήσει έχουν να κάνουν με το νομοθετικό και υποπτικό τμήμα. Πάντω, ένα πω ότι και εμείς ε, ως ε, αρχή εξυγίανσης ε, εξετάζουμε τους ομίλους στο σύνολό τους. Εάν δηλαδή υπάρχουν κάποια στοιχεία του ομίλου σε μαύρη λίστα θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και θα πρέπει να εξετάζουμε τον όμιλο στο σύνολό του λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία. Η εξυγίανση της εγκατάστασης σε χώρα μαύρης λίστας, αυτό είναι θέμα των ε, χωρίων αρχών, αλλά βέβαια πρέπει να εξετάζουμε στο σύνολό του τον ε, όμιλο. Ε, ο κύριος Ζήλε, σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας μιλάει ε, από τη θέση που έχει και σύμφωνα με το ισχύον ε, νομικό πλαίσιο. Αλλά πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε επιθυμίες για το τι θα θέλατε να αλλάξει ε, και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω Ε, τον κύριο Γιάννα που αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο που δημιουργεί κάποιες αβεβαιότητες. Υπάρχουν τράπεζες ε, σε μικρά κράτη-μέλη που δεν ε, εποπτεύονται από τη Φραγκφούρτη και σε μικρά κράτη-μέλη αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες δυσκολίες. Ίσως θα μπορούσε λοιπόν ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός ή η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ε, να βοηθήσει τις τράπεζες αυτές ε, με την αδειοδότηση σε κρίσιμες περιπτώσεις. Όσον αφορά την ε, καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων, έχουμε και την προληπτική εποπτεία. θα διαπιστώσετε ότι οι δείχτες είναι εντάξει για ε, του, τις τράπεζες αυτές, αλλά Εάν όλοι οι δείκτες ε, είναι εντάξει, ε, μπορεί παρόλα αυτά να μην έχουμε ε, στοιχεία για την νομοποίηση παράνομων εσόδων για τις τράπεζες αυτές. Και Ρωτήσατε ποια κράτη-μέλη έχουν προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή όσον αφορά τους αλλοδαπούς καταθέτες. Ε, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει, διότι υπάρχουν πολύ μικρά κράτη-μέλη με πολύ καλή γνώση του τραπεζικού τομέα, με ελάχιστες ε, ποινικέ ε, υποθέσεις που δεν μπορούν να λάβουν ε, τις σωστές αποφάσεις. Ε, νομίζω κάτι στραβό υπάρχει στο σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. like Mr. Σας ευχαριστώ. Ποιος θα θέλει να ξεκινήσει. Ο κύριος Χάμπεν, παρακαλώ. Ε, όσον αφορά τον ε, κατάλογο των χωρών. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω αργότερα αφού μιλήσω με τους νομικούς μου, αλλά αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι μερικές φορές μιλάμε για την πρόκληση όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν είναι επειδή δεν νοιάζονται οι διάφοροι άνθρωποι, μπορεί να είναι επειδή υπάρχει ε, εθνική νομοθεσία που εμποδίζει το μοίρασμα των πληροφοριών. Σε έναν κόσμο λοιπόν όπου με μια οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης, ε, εάν υπάρχουν ε, εθνικοί κανόνες ε, για που να απαγορεύει την ανταλλαγή δεδομένων, αυτό δεν θα βοηθήσει τους ανθρώπους στη μονάδα χρηματοπιστωτικών πληροφοριών να στείλουν πληροφορίες στους επόπτες θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση με τις κατευθυντήρες γραμμές και να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν εμπόδια όσο θα έχουμε το νομικό πλαίσιο που έχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκράντε. Να πω στον κύριο Τσίλε ότι Όσον αφορά την ανάγκη να επιδιώξουμε την σύγκληση, αυτό ισχύει όχι μόνο για τις αρχές της Τραπεζικής Ένωσης, ε, αλλά και για τις μικρές τράπεζες που ε, προς το παρόν ε, παραμένουν ευθύνη των εθνικών αρχών. Έχουμε λοιπόν τις τράπεζες σε πτώχευση ή πιθανή πτώχευση. Ε, στις περιπτώσεις αυτές είναι ακόμα πιο σημαντικό διότι ε, είναι πιθανότερο να διαλυθούν παρά να εξηγενθούν οι πολύ μικρές τράπεζες. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε προς ένα πλαίσιο όπου να μπορέσουμε να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα για τις τράπεζες σε κεντρικό φορέα. για μας ισχύει, αλλά νομίζω ότι και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ισχύει ότι ε, οι μοιρασμένε αρμοδιότητες ίσως να μην, να λειτουργούν πολύ καλά στην πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σουγιάννα. Κάτι που νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε τώρα που μας ζητάτε να εκφράσουμε επιθυμίες. Αναφέρθηκε πριν ε, ότι θα είναι χρήσιμες οι αξιολογήσεις, ε, οι ικανότητες και αυτό συνδέεται με θέματα νομοποίησης παράνομων εσόδων. διότι μπορεί με αυτή τη βάση να καθοριστεί η ικανότητα μιας τράπεζας ή η ανικανότητά της. Υπάρχουν κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν μεταφερθεί με πολύ διαφορετικό τρόπο στις ε, διάφορες ε, χώρες και πολύ συχνά μόνο ε, ποινικέ αποφάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις κεντρικές αρχές και τέτοιες διαφορές δημιουργούν σημαντικά προβλήματα για μας στη δουλειά μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας θυμίσω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ κύριε Τόρβαλτς της Ευχαριστώ. Αφού άκουσα τους συνήθεις ύποπτους στο πρώτο πάνελ, μου έκαναν εντύπωση οι 72 και 17 σελίδες που ανέφερε ο κύριος Κόλσον, γιατί δεν ξέρω αν ε, ε, σωστά κατευθυνόμαστε. Αν μπορούμε να εντοπίσουμε κάπως ε, τις οδηγίες σας, θα πρέπει να ακούσουμε και τον κόδωνα κινδύνου ή θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο, γιατί από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα είναι πολιτικά, δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είναι, είναι δικό σας πρόβλημα, λένε όλοι. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να δούμε πού μπορεί να, να, να ορθωθούν εμπόδια, μήπως πού δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε περισσότερο. Γιατί πρέπει να λύσουμε και τα πολιτικά προβλήματα και αυτό είναι ο τρόπος που πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Άμπανα ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και για τις κατευθυντήριες γραμμές. Ε, όντως αξίζει τον κόπο να ε, τις ερμηνεύσουμε. Ναι, έχουμε κατευθυντήριες γραμμές, αυτό λέτε. Εφόσον όμως κανείς δεν τις χρησιμοποιεί, τότε τι νόημα έχει. Πάντως, αν υπάρχει ένα πράγμα που μπορούμε να καταφέρουμε χωρίς να αλλάξουμε την νομοθεσία είναι ανεξάρτητες ε, ε, εκθέσεις δεν υπάρχει εκεί παραβίαση της ε, κοινοτικής νομοθεσίας. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε εκεί με τις αρμόδιες αρχές, να εντοπίσουμε τομείς όπου ε, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, χρησιμοποιούνται οι κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό ίσως κάτι θα προσέθετε. Κάπως αρχίσαμε να κινούμαστε προς τη ζεστή κατεύθυνση. Δεν θα γίνονταν όλα τέλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, τι μπορούμε να κάνουμε για τις κατευθύνσεις γραμμές εφόσον ο κόσμος δεν τις ακολουθεί, ε, θα μπορούσαμε ίσως να δουλέψουμε με τους συναδέλφους στις αρμόδιες αρχές. Κάτι θα προσέφερε αυτό. Σας ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις? Όχι. Είστε ευχαριστημένοι λοιπόν. Ωραία. Οπότε τώρα πάμε στους πράσινους. η Εύα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ έχω μια ερώτηση για τον κύριο Χάμπον. Για σας ναι. Μετά από το σκάνδαλο του Παναμά, εσείς ε, νομίζω ζητήσατε από τις εθνικές αρχές, ρωτήσατε μάλλον τις εθνικές αρχές, τι έχουν κάνει τι σκοπεύουν να κάνουν για να παρεμποδίσουν την εμφάνιση νέων ε, σκανδάλων τύπου Παναμά. Μας είπατε ότι τρεις χώρες είπαν πως δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι σημαντικό η Επιτροπή μας να γνωρίζει ποιες ήταν αυτές οι τρεις χώρες ε, και για ποιους λόγους δεν έκαναν τίποτα. Εμείς ακούσαμε τις αρχές της Μάλτας να λένε ότι ήθελαν κατευθυντήριες γραμμές και καταλαβαίνω πως έχετε φτιάξει κάποιες. Οι κατευθυντήριες σας γραμμές ε, αξιολογούν και ποιος είναι και ο κατάλληλος για να είναι κεφαλής της τράπεζας και πιστεύετε ο κύριος Άλισάντερ θα είχε ε, θα, θα τηρούσε τις προϋποθέσεις για να είναι επικεφαλής της τράπεζας. Μπορεί κανείς να διοικήσει μια τράπεζα με 130 πελάτες όπου η μισή εξ αυτών όπου η μισή είναι ανύπαρκτη. Και πώ θα λειτουργήσουν οι εθνικέ αρχέ υπ' αυτέ τι θετικέ, όταν ξέρουμε πω ο ίδιο ο Πρωθυπουργό πήγε στη γάμο αυτού του κυρίου το Κοινοβούλιο συχνά έχει ζητήσει κεντρική μονάδα για την ε, σε χρηματοπιστωτικές πληροφορίες. Ε, ε, εσείς πιστεύετε πως θα ήταν θετικό να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό FIU ή πιστεύετε πως η συνεργασία είναι καλύτερος τρόπος και αν είχαμε ευρωπαϊκή FIU, τι μορφή θα είχε. Να απαντήσω ευχαρίστω. Λοιπόν, έγινε μία έρευνα για το αν τα πράγματα ήταν τέλεια και αν πράγματι επειδή ήταν τέλεια δεν είχαν υπάρξει αλλαγές. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε όμως να δώσουμε ονόματα σε σχέση με τις συγκεκριμένες χώρες. Οι κατευθυντήριες γραμμές ε, βασίζονται στην αξιολόγηση των κινδύνων και στον εντοπισμό των πιθανών κινδύνων. Όταν βλέπει κανείς τα παγκόσμια ε, επίπεδα στάνταρτ, βλέπει ότι έχουμε ε, κάποιους δεσμούς στην Ευρώπη μεταξύ μας σε επίπεδο αρχών που ασχολούνται με το φαινόμενο, αλλά ίσως ασθενών δεσμών. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί αυτοί. Τώρα, αν περιμένει να καταδικαστεί πλήρως και να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταδίκης κάποιου σε ποινικό επίπεδο, αυτό είναι κάτι το οποίο άπτεται του εθνικού δικαίου και συνήθως είναι ιδιαίτερος χρονοβόρο. Μπορεί να απαντήσει λοιπόν κανείς διπλά. Πρώτον, κατευθυντήριες γραμμές με διαφορετικό τρόπο και ίσως οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές να συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύτερα. σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε, αν οι ρυθμίσεις είναι οι κατάλληλες. Τώρα, ε, για τη συλλογή χρηματοπιστωτικών πληροφοριών. Εμείς δεν είμαστε η Financial Intelligence Unit. Πιστεύουμε ότι η συλλογή των πληροφοριών και η διανομή των πληροφοριών και η αμοιβαία ανταλλαγή των πληροφοριών είναι κάτι το χρήσιμο. Εμείς αναλύουμε επίσης δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για άλλα θέματα, όπως οι δοκιμασίες των τραπεζών. Δεν είναι δική μας δηλαδή αρμοδιότητα να πούμε αν μια τέτοια υπηρεσία συλλογής χρηματοπιστωτικών πληροφοριών θα ήταν καλή ή όχι. Για την ΚΟΕ. Θα ήθελα καταρχάς να ρωτήσω το εξής. Από τη μία μεριά το πρώτο πάνελ έδειξε πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα ε, στην Ευρώπη και το δεύτερο πάνελ έδειξε επίσης τι προβλήματα υπάρχουν. Ε, διάφοροι ύποπτοι αναφέρθηκαν ήδη. Εγώ θα ήθελα να κοιτάξουμε λίγο την Γερμανία. Ξέρουμε ότι στη χώρα μας ε, Υπάρχουν σημαντικέ ελλείψει όσον αφορά την καταπολέμηση τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Το 78% των υποθέσεων ε, είναι δύσκολο να παρακολουθούν στη συνέχεια. Και τι μπορούμε να κάνουμε. προ τον κύριο Χάμπεν, την τελευταία εβδομάδα το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο Υιοθέτησε την πέμπτη οδηγία για την ε, καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Ε, η ομάδα μου επικροτεί το βήμα αυτό του Κοινοβουλίου. Από την άλλη δεν καταφέραμε καμιά τεράστια αλλαγή εσείς. Πώς βλέπετε την οδηγία αυτή και πώς βλέπετε τις δυνατότητες ε, επιβολής κυρώσεων αρκούν Επίσης, όσον αφορά την σχέση του, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής με τις Εθνικές Αρχές, για παράδειγμα τη Γερμανία, αυτή τη στιγμή όλες οι εθνικές αρχές δείχνουν ιδιαίτερο ίστρο για την ε, εφαρμογή των κανόνων. Πώς ε, αξιολογείτε εσείς τις δυνατότητες να γίνει αυτό. Και τέλος, ε, προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί που σας εμποδίζουν ε, να ε, καταπολεμήσετε επαρκώς την νομοποίηση παράνομων εσόδων. Ε, πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες του, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Σας ευχαριστώ κύριος Χάμπεν. Well, thank you for the... Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Πολύ λογικές. Όσον αφορά την πέμπτη οδηγία και τις κυρώσεις, αρκούν οι κυρώσεις. Το θέμα δεν είναι ποια είναι η πιο ε, αυστηρή ποινή που μπορεί να επιβληθεί. Πιο πολύ με απασχολεί η συνεπής ε, και σωστή εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο από το να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια νέα σκληρότερη ποινή. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα την ερώτηση ανάμεσα στο, ε, ε, για το θέμα, ε, για τη σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και στις Εθνικές Αρχές. Ε, ναι, η ερώτησή μου ήταν, μπορείτε να διασφαλίσετε οι εθνικές αρχές να μπορούν να πληρούν καλύτερα τα καθήκοντά τους. Με απλά λόγια στο ισχύον πλαίσιο υπάρχουν περιορισμοί στην ε, δυνατότητα να υποπτεύουμε τις ε, εθνικές αρχές. Δεν είμαστε επόπτης, ούτε μπορούμε να τους πούμε πώς να κάνουμε τη δουλειά τους. Ε, εάν δεν ακολουθούν τους κανόνες, τότε μπορούμε να επισημάνουμε την παραβίαση. Οι αξιολογήσεις ομοτήμων λειτουργούν πολύ καλά στην πράξη, αλλά όταν έχουμε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που δείχνουν τι πρακτικές χρησιμοποιούν και αξιολογούν ένα τον άλλον τελικά καταλήγουμε στο τι είναι καλό, καταλήγουμε ποιες είναι οι μεγάλες ε, ανομαλίες που υπάρχουν στο σύστημα, αλλά δεν ε, υπάρχει τρόπος ε, για εναρμόνιση. Πιστεύουμε ότι οι αξιολογήσεις ομοτήμων μπορούν να δώσουν πολύ καλή και λογική κριτική και σκληρή κριτική στο ισχύον πλαίσιο. Αλλά βέβαια κάτι τέτοιο απαιτεί και κάποια νομική τροποποίηση αλλά και επαρκείς πόρους. Ε, ναι, παρακαλώ είστε σύντομος διότι είναι περιορισμένος ο χρόνος μας. Ναι, σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι η αρμόδια αρχή για θέματα νομοποίησης παράνομων εσόδων. Το ρόλο μας εδώ λοιπόν το βλέπουμε ως εξής Τα ευρήματα στον τομέα της νομοποίησης παράνομων εσόδων που έχουν ανακαλύψει οι εθνικές αρχές, αυτά φροντίζουμε να αντικατοπτρίζονται στην ε, εποπτική μας αξιολόγηση. Ε, διότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε τον κίνδυνο για τις ε, τράπεζες αυτές και το είδαμε τη σημασία αυτών των κινδύνων στην περίπτωση της τράπεζας ABLB. Μπορεί να υπάρχουν επίσης κίνδυνοι λόγω των κίνδυνοι στη συνεργασία λόγω των προστήμων, μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι για τη διακυβέρνηση, εφόσον γίνει γνωστό ότι χρησιμοποιείται για την νομοποίηση παρανομών εσόδων η τράπεζα. Ο βασικός περιορισμός μας είναι ότι μερικές φορές δεν έχουμε τις πληροφορίες για να μπορούμε να τις αντικατοπτρίσουμε στην αξιολόγησή μας. Μερικές φορές μπορεί να συναντούμε κάποιες ελλείψεις, για παράδειγμα στις επιτόπου επιθεωρήσεις μπορεί να ανακαλύψουμε κάποια στοιχεία ε, έλλειψης ε, όσον αφορά τους ελέγχους για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων στην τράπεζα. Αλλά δεν είμαστε η αρμόδια αρχή και χρειαζόμαστε πληροφορίες από την αρχή που είναι αρμόδια για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Δεν ε, ε, πρέπει λοιπόν να μπορούμε να βασιζόμαστε σε έγκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριος Φάντεν Κεντελάρη, θα ήθελα να θέσω στα Ολλανδικά την ε, ερώτησή μου. Ε, πώς μπορούμε να έχουμε συστήματα συναγερμού. Η Ευρωπαϊκή η Διερευνητική Επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά είπε ότι οι άδειε των τραπεζών είναι σημαντικέ, μπορούν να ανακληθούν. Ε, χρειαζόμαστε σαφείς κυρώσεις για τράπεζες ε, που κάνουν ε, επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Θα πρέπει να ε, εμποδίσουμε τις δραστηριότητες αυτές, θα πρέπει να ανακαλούνται οι άδειε των τραπεζών αυτών, εφόσον δεν τηρεί κανείς τους κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε ότι δεν είναι αρμόδια για θέματα νομοποίησης παράνομων εσόδων, αλλά ε, έχει το εργαλείο των αδειών των, των τραπεζών. Είδαμε ε, στις περιπτώσεις των εγγραφών του Παναμά ε, ανάκληση αδειών τραπεζών και είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για μικρές τράπεζες ε, που μπορεί να έχουν επιπτώσεις και σε αλλα κρατημέλη. Σήμερα το πρωί υπόθηκε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα μέχρι να φτάσουμε σε έναν ενιαίο μηχανισμό στην Ευρώπη για να ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά. Ίσως θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε μια διάμεση λύση. Αναρωτιέμαι για παράδειγμα αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τα stress test για να κάνει τέτοιους ελέγχους να έχουμε και ένα σύστημα συναγερμού. Το stress test, ε, ε, το τεστ προσωμείωσης ακραίων καταστάσεων μπορεί να γίνει και τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν για να ε, χτυπήσουμε συναγερμό. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εάν αυτό είναι απαραίτητο, μπορεί να ανακαλέσει τις άδειες ή να ζητήσει την ανάκλησή τους. Έχουμε παραδείγματα όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει κάνει τίποτα. Γιατί? Ο κύριο Σουχένα, σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, όταν αφορά την αφαίρεση της, άδειας, ε, της τραπεζικής άδειας, θα ήθελα να διευκρινίσω πως όντως, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, υπάρχει υπάρχει βάση για αφαίρεση της άδειας λόγω των διατάξεων περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης παρανόμου προσόδων. Προβλέπετε Τώρα πώς πάει στην πράξη στο SSM, είμαστε αρμόδια αρχή για να αποσύρουμε την, άδεια, την τραπεζική άδεια, αλλά αν η μόνη βάση για την αφαίρεση της άδεια σχετίζεται στην ε, ξέπλυμα χρήματος, επειδή δεν είμαστε εμεί αρμόδιοι γι' αυτό, χρειάζονται και πάλι πληροφορίες που προέρχονται από τις ε, αρχές ε, AML για να μπορέσουμε να προβούμε στην αφαίρεση της άδεια. Έχουμε παραδείγματα στο παρελθόν που το έχουμε κάνει αυτό. Αλλά και πάλι πρέπει να βασιστούμε στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις αρμόδιες αρχές και βεβαίως θα πρέπει η παράβαση να είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι, μήνυμα, δεν είναι κάποιες ελάχιστες ε, παραβάσεις. Είναι το, απότε, το ίστατο μέσο, ίστατη κύρωση αυτή. Και άρα πρέπει να χρησιμοποιείτε φρόνημα και συνετά. Τώρα, πώς, πώς εντοπίζουμε τους κινδύνους AML σας εξήγησα πώς κάνουμε τις εκθέσεις μας, ε, τη δυνατότητα να το, να το συμπεριλάβουμε στο, στις δοκιμές Αυτό ίσως θα πρέπει να το αναπτύξουμε περισσότερο. Πάντως ε, δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα τέτοιο παλιότερα, αλλά ότι στο ευρύτερο πλαίσιο της ιδιαιτερότητας αυτών των stress test αναλύουμε το επιχειρηματικό μοντέλο και αν ανακαλύψουμε πως το, αυτό το μοντέλο είναι επικίνδυνο λόγω για παράδειγμα της αναλογίας των ε, λοδαπών ε, πελατών τότε αυτό που κάνουμε είναι επιβάλλουμε επιπλέον απαιτήσει ρευστότητα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η τράπεζα θα είναι πιο ανθεκτική σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Ήδη το κάνουμε αυτό, αλλά μετά από την υπόθεση EVLV και τις άλλες που αναφέρθηκαν σήμερα το πρωί, ε, σκεφτόμαστε για τη μεθοδολογία μας πώς θα την ενισχύσουμε περισσότερο ώστε να καλύψουμε τέτοιου είδους κινδύνους. Και για την αφαίρεση της άδεια, όπως είπα πριν, μπορούμε να αφαιρέσουμε την άδεια, αλλά η αφαίρεση της άδεια ε, σχετίζεται μόνο με EML Χρειαζόμαστε επιβεβαίωση των σχετικών πληροφοριών και ειδικά για τις υποθέσεις που συζητήθηκαν σήμερα το πρωί. Η ΕΚΤ έχει αναμειχθεί, αλλά και όπου δεν έχει ακόμα αφαιρεθεί άδεια, σημαίνει ότι ασχολούμαστε με τις αθηνικές αρχές να δούμε αν πρέπει να αφαιρεθεί ή όχι. Δηλαδή η διαδικασία είναι υπό εξέλιξη σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι ένα Αγγίλ, από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που είναι σαφές μετά από τη συζήτηση που προηγήθηκε είναι ότι ανάγκη υπάρχει για μεγαλύτερη συνεργασία. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν και κάποιοι έμεσοι τρόποι καλύτερη συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Transparency International είπε ότι υπάρχουν 4,4 δις βρετανικής ιδιοκτησίας ύποπτα κεφάλαια, ύποπτες αποδείξεις πλούτου. Ε, δεν έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα απέναντι και σε ρωσικές εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται οι συναλλαγές ε, με τους Ρώσους έχουν συνεχιστεί και ένας από τους τρόπους που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό είναι και μέσω του ΣΥΤΙ. Οι Ρώσοι εξακολουθούν να μπορούν να δανείζονται και αφού παίρνουν τα χρήματα αυτά μπορούν να τα δίδουν στις τράπεζες οι οποίες με τη σειρά τους υφίστανται τις κυρώσεις. Αυτό λοιπόν θα ήταν ε, ένας από τους χώρους, ένας από τους τρόπους έτσι ώστε να προσπαθήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συντονιστούμε. Επίσης αναφέρομαι και σε αυτά τα οποία λέτε στα γραπτά σας. Λέτε ότι ε, για συγκεκριμένες ε, ε, ενέργειες είσαστε σε θέση να αναλάβετε δράση και σε ποια στιγμή ε, είναι αν θέλετε η κρίση, ποια στιγμή είναι η κρίσιμη στιγμή όπου η τράπεζα αποφασίζει ότι θα εμπλακεί σε μια διαδικασία και ότι έχει τα κατάλληλα μέσα για να το κάνει. Αυτή είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται και για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος, ιδιαίτερα μετά από ενημέρωση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Και σαν ελεγκτή των συστημικά σημαντικών τραπεζών, αξιολογείται τους κινδύνους και οι περιπτώσεις που συζητήσαμε σήμερα δείχνουν ότι οι τράπεζες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν σκάνδαλα με την TSB και άλλες τράπεζες. Ε, υπάρχουν προβλήματα με τα πληροφορικά του συστήματα. Αν δεν πάνε καλά τα πληροφορικά συστήματα, παίρνετε κυρώσεις εις βάρος τους. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις Υπάρχουν θέματα στα οποία δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις στην παρούσα φάση, αν και χρήζουν περαιτέρω έρευνας. θα μπορούσε να δημιουργηθούν αν αφήσουμε ανεξέλεκτα τα πράγματα πάρα πολλές παρενέργειες. Σχετικά με την καθημερινή μας πρακτική στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμείς ε, κάθε πότε ε, προχωράμε στις αξιολογήσεις αυτό που λέμε fit and proper. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιους αξιολογήσεις ε, για τις συστημικές τράπεζες, όπως επίσης και για τους διαχειριστές των πιστοτικών ιδρυμάτων, όχι για τους μετόχους κυρίους ή όχι. και όταν θέλουν ας πούμε οι τράπεζες να ορίσουν ένα νέο υψηλού επίπεδου στέλεχος προφανώς και εκεί μπορούμε να ζητήσουμε ενημέρωση αλλά η ευθύνη έγκυται φυσικά στο ίδιο το πιστοτικό ίδρυμα. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για να αξιολογήσουν την ποιότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα. Εμείς κάνουμε μία πρώτη αξιολόγηση και αν τυχόν δούμε ότι υπάρχουν κάποια συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν εμπόδια στις πιστοτικές δραστηριότητες, τότε παρεμβαίνουμε εκ νέου. Δεν παρεμβαίνουμε δηλαδή σε τακτική βάση, κάνουμε την πρώτη αξιολόγηση βέβαια, αλλά αν κάποιες από τις συνθήκες, κάποιες από τις προϋποθέσεις τις οποίες είχαμε επιβεβαιώσει στην πρώτη αξιολόγηση δεν ισχύουν πλέον, τότε παρεμβαίνουμε εκ νέου. πόσες ε, αφαιρέσεις άδεια λειτουργίας είχαμε μέχρι τώρα μετά από παραβιάσεις του κανονισμού για ξέπλυμα. Δεν είναι πολλές. Έχω δύο ε, περιπτώσεις στο μυαλό μου και μία τρίτη. Και δεν θα, ε, αναφερθώ σε ονόματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξουν δύο με τρεις τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα τι κάνουμε με τους λειτουργικούς κινδύνους και τις αδυναμίες των πληροφορικών συστημάτων. Προφανώς και τα αξιολογούμε και τις δυνατότητες και ικανότητες που έχουν σε μια τράπεζα. Άμα δούμε ότι το προφίλ της τράπεζας παραμορφώνεται ή αποδυναμώνεται λόγω των ελλείψεων στον τομέα των πληροφορικής, των ηλεκτρονικών, τότε ζητάμε από την τράπεζα να, υπο, υποβάλει ένα πρόγραμμα το οποίο θα τη βοηθήσει να ξεπεράσει τις αδυναμίες αυτές. Και αν θεωρήσουμε ότι λόγω αυτών των αδυναμιών οι κίνδυνοι τους οποίους εκτίθεται η τράπεζα είναι υψηλοί, τότε ε, φυσικά παρεμβαίνουμε πάλι έτσι ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα της τράπεζας να αντέξει σε τέτοιου είδους θέματα, προβλήματα. Η Άννα Γκόμες ήθελε τον λόγο στα πλαίσια του Κατστιάη, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γι' αυτό διμερώς θα μπορέσετε να θέσετε την ερώτησή σας ή γραπτά. Πριν ευχαριστήσω τους ομιλητές μας θα ήθελα να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Είναι σαφές, έχει, ε, πλέον είναι φανερό και έχει επιβεβαιωθεί ότι σε ορισμένες χώρες οι αρχές παρακολούθησης και εποπτείας λειτουργούν αλλά η συνεργασία μαζί τους είναι ανεπαρκής. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει, αυτό είναι σαφές. Υπάρχει χώρος για συγκεντρωτικότερα συστήματα. Κάποιοι θέλουν ε, τα συστήματα αυτά να λειτουργούν κυρίως σε εθνικό επίπεδο, κάποιοι όχι. Κάποιοι ζητούν επίσης να υπάρξει μια ευρωπαϊκή αρμόδια αρχή για το ξέπλυμα. και βλέπουμε ότι οι οικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται από τις ε, αρμόδιες αρχές δεν επιτρέπουν υποχρεωτικά τον εντοπισμό των κινδύνων ε, για ξέπλυμα χρήματος. Έχουμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες όπως στην περίπτωση της Λετονικής Τράπεζας αλλά συνολικά μπορούμε να πούμε ότι πολλοί πιστεύουν ότι έχουμε ίσως αρκετά καθυστερήσει, αλλά απαιτείται να υπάρξει καλύτερος ευρωπαϊκός συντονισμός και ίσως και μια κεντρική ευρωπαϊκή υπηρεσία. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους τους ομιλητές, εκτιμώ την παρουσία σας και τις απαντήσεις σας.